Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ζητώ συγγνώμη που αρχίζουμε με μια καθυστέρηση πέντε λεπτών. Αλλά κάπως χάθηκα. Πήγα σε, σε, σε λάθος συνεδρίαση, γιατί σήμερα συνεδριάζουμε αλλού. Μια που αναζητούμε πάντα το καινούριο, ζητούμε και νέους αίθουσες. Σας χαιρετίζω όλους, σας καλημερίζω. Θα ήθελα να σας πω, θα ξεκινήσουμε με την μήνυα ακρόαση για το πρόγραμμα δράσης. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με, το, με τη γραφειοκρατία. Ένα θέμα που διατυπώθηκε ήδη τον τελευταίο καιρό και η συνάδελφος στην είχε δικαίως τονίσει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Γι' αυτό καλέσαμε κάποιους ενδιαφέροντες εμπειρογνώμονε υψηλωτά του επίπεδου και ελπίζουμε να ακούσουμε πολλά καινούρια πράγματα. Μία μικρή παράκληση εισαγωγικά. Παρακαλώ να τηρήσετε όλοι το χρόνο ομιλία που έχει συμβοληθεί. Γιατί αλλιώ έχουμε τεράστιο πρόβλημα να ολοκληρώσουμε τι εργασίε μα σήμερα. Αυτό σημαίνει οι εμπειρογνώμονε να μιλήσουν με ακρίβεια να παρουσιάσουν απόψεις τους και οι συνάδελφοι στο δεύτερο γύρο στις ερωτήσεις τους να δείξουν κάποια εγκράτια. Χθε είχαμε προβλήματα να τελειώσουμε έγκαιρα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα Κρίστοφερ Χάλερ που θα μας κάνει μια παρουσίαση από τη σκοπιά της ερευνητική κοινότητα. Παρακαλώ. Thank you very much, Chairman. members of Parliament. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος πλαίσιο. Ε, υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα, προβλήματα τα οποία πραγματικά πρέπει επιγόντως να λάβετε υπόψη σας και θέλω να ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα βρει ικανοποιητικές λύσεις. Μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν προβλήματα μετάφραση τη διερμηνία. Υπάρχουν ίσω κάποιε καμπίνες που δεν ακούγονται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό παρακαλώ. Oder betrifft das nur die deutsche Kabine? Only the German translation? Dann mache ich das auf Deutsch. Dann verstehen die anderen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 Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, υπάρχει ένα πρόβλημα ναι. μόνο στη γερμανική διερμηνία, μόνο στους διερμηνείς, στην, τεχνολογική. τεχνική. Ε, να ακούσουμε τι θα πείτε στα αγγλικά κατευθείαν. Και όποιοι θέλουν να τα ακούσουν στα γερμανικά, ας περιμένουν 2-3 λεπτά, θα διορθωθεί. Χρειάζεται λίγο χρόνο. Συμφωνείτε? Ωραία. Ξανά, κύριε Χόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου που με καλέσατε σήμερα και θα προσπαθήσω να μιλάω καθαρά ε, στην περίπτωση που τελικά ε, δεν μπορεί να μεταδοθεί η γερμανική διερμηνία. Λοιπόν, να σας περιγράψω καταρχήν τους ε, οργανισμούς που εκπροσωπώ. Ίσως έτσι θα καταλάβετε καλύτερα αυτό που θέλω να σας πω. Έχουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανώσεων Έρευνας και Τεχνολογία. Το ακρονίμιο είναι EARTU, o, με συγχωρείτε, o. Είναι περίπου 150 οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεμένες χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτή την ομοσπονδία. Το ERTO τι ακριβώς είναι, να το πω πιο απλά. Πρόκειται για οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας ε, ε, που ε, χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, άλλες πάλι είναι καθαρά κρατικές και η βασική τους αποστολή είναι να έρθουν αντιμέτωποι με τα βασικά θέματα, τις βασικές προκλήσεις ε, της σημερινής εποχής, όπως επίσης και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα. Σύντομα θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τις ε, πιο μεγάλες και γνωστές οργανώσεις, ξεκινώντας από το βορρά προς το νότο της Ευρώπης, αλλά θα συμπεριλάβω και οργανισμούς όπως VTT στη Φίνδα ή Σύντεφ στην Νορβηγία, ε, τα περισσότερα βιομηχανικά Ινστιτούτα στη Σουηδία, το Δανικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο στη Δανία, Γερμανία, την TAO στην Ολλανδία, VNO στο Βέλγιο, ε, στην Γερμανία έχουμε οργανώσει σε τεχνολογικούς εταίρου και ιδρύματα στην Πολωνία, το Institute Carnot στη Γαλλία, τα τεχνολογικά κέντρα στην Ισπανία και πάρα πολλού άλλου. Οι οργανισμοί έρευνας και τεχνολογία είναι πολύ σημαντικοί στο πρόγραμμα πλαίσιο. Ο γερμανικός οργανισμός Fraunhofer είναι ο δεύτερος ε, μεγαλύτερος ιδιώτης ε, εταίρος ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 6. Οι πέντε μεγαλύτεροι οργανισμοί έρευνας και τεχνολογία που σας ανέφερα από κοινού εκτέλεσαν 1.400 προγράμματα στο πρόγραμμα πλαίσιο 6 μιλάμε για περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μη πανεπιστημιακοί οργανισμοί έρευνας είναι περίπου το 1 τρίτο, έλαβαν το 1 τρίτο της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα πλαίσιο Περθμών 6. Πρόκειται για ένα σημαντικό τομέα. Και κάτι στο τέλος, εν είδη εισαγωγής, Πολύ συχνά ακούμε ότι το πρόγραμμα πλαίσιο είναι το 5% των δημοσίων κονδυλίων για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ευρώπη. Σωστό αυτό, αλλά ο αριθμός αυτός δεν αποδίδει την πραγματική σημασία του προγράμματος πλαίσιο. Θα πρέπει να έχετε πάντα κατά νου ότι τα κρατικά κονδύλια για την έρευνα και την τεχνολογία καλύπτουν και κονδύλια για την υποδομή, για την ανέγερση πανεπιστημίων και επίση καλύπτουν και βασικούς μισθούς που καταβάλλονται σε πανεπιστημιακούς δασκάλους και σε άλλους ερευνητικού φορείς. Αν λοιπόν προσπαθήσει κανείς να καταργήσει αυτά τα κονδύλια, θα πρέπει να έχει κυρίως κατά νου ότι μιλάμε για ε, κονδύλια που χορηγούνται σε συγκεκριμένα και σημαντικά προγράμματα. Το πρόγραμμα πλαίσιο είναι περίπου το 25% του συνόλου της ε, επιδότησης ε, από κρατικής πλευράς για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Αυτό είναι σημαντικό γιατί καταδεικνύει την μόχλευση ε, που μπορεί να ε, προκαλέσει η έρευνα και η τεχνολογία στην Ευρώπη. Και το δεύτερο που πρέπει κανείς να έχει κατά νου είναι το πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι το μόνο σημαντικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας που στηρίζει διασυνοριακά υπερεθνικά προγράμματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Άρα δηλαδή το πρόγραμμα πλαίσιο για αυτούς τους λόγους πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Θα έρθω λοιπόν τώρα στα θέματα που θα εξετάσουμε σήμερα. Θα μπορούσα να σας αναφέρω ένα μακρύ κατάλογο προβλημάτων, αλλά δεν θέλω να εμπλακώ σε τεχνικής ε, φύσης ε, λεπτομέρειες. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές βελτιώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που είναι το αποτέλεσμα πόντων συστημικών προβλημάτων που αν δεν λυθούν αυτά δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ε, πρόοδος. Και αυτό είναι το θέμα που θέλω να εξετάσω σήμερα. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα πλαίσιο 7 είχε ως στόχο να επιφέρει σημαντικές ε, γραφειοκρατικές απλουστεύσεις. Να αναφέρω ορισμένα. Υπήρξαν ε, σημαντικές βελτιώσεις και θα ήθελα να φέρω εδώ παραδείγματος χάρη την δυνατότητα μίας και μόνο καταγραφής, τα διοικητικά εργαλεία που εισήχθησαν ή αν θέλετε την σύσταση των εκτελεστικών φορέων. Όλα αυτά με την πάροδο του χρόνου θα δείξουν ότι αποτελούν <clears throat> πολύτιμες βελτιώσεις. Υπάρχουν και κάποιες άλλες απλουστεύσεις που ήδη έχουν εφαρμοστεί εν μέρη, που δεν είναι βέβαια τόσο ευχάριστες και μάλιστα μερικές εξ αυτών ε, θεωρούνται και αποτυχία. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ε, θα αναφερθώ στο θέμα των εφάπαξ ποσών, ε, του ενιαίου κόστου στα πάγια, σταθερά ποσά. Στα αποκαλέσουμε έτσι χάρη της ε, ευκολίας. Αυτά προτάθηκαν ε, ως απλούστευση, ίσως και να αποτελούν κάποια απλούστευση για την Κομισιόν, όμως δεν είναι απλούστευση ούτε καν διευκόλυνση για τους περισσότερους που συμμετέχουν στα προγράμματα πλαίσιο. Είτε είναι είτε λιγότερο, είτε είναι μεγάλοι είτε λιγότερο μεγάλοι οργανισμοί. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα σύστημα λογιστικό που, καλύπτουν, που καλύπτει όλα τα, όλες τις δαπάνες. Όταν ας πούμε κάποιος ε, συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα, παίρνει το αεροπλάνο, μένει σε ξενοδοχείο, το κόστος εντάσσεται στο λογιστικό σύστημα, στο πραγματικό κόστος, στο πραγματικό ποσό που καταβάλλεται. Και όταν η Κομισιόν επιστρέφει το ποσό στον ενδιαφερόμενο, ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο όμως δεν ε, αντικατοπτρίζει τις δαπάνες, δεν έχει σχέση με τις δαπάνες που έγιναν, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Άρα δηλαδή εδώ προκύπτει επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Ίσως να μην σας φαίνεται τόσο σημαντικό, αλλά οπωσδήποτε εδώ δεν πρόκειται για απλούστευση για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ υπάρχει και κάποιος κίνδυνος, γιατί υπάρχει, ασκείται πολιτική πίεση από εκείνου ε, που δεν θέλουν να υπάρχει διασπάθηση του κρατικού χρήματος ή να υπάρχει ε, περιθώριο για εκμετάλλευση από πλευράς ιδιωτών. Άρα δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και ε, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στην ε, πραγματικά παράδοξη κατάσταση που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα για το πρόγραμμα Marie Curie στο πρόγραμμα πλαίσιο 6 όπου είχαμε φάπαξ ποσά, οι ελεγκτές ε, ζήτησαν αποδείξεις ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για ένα συγκεκριμένο θέμα ήταν ε, τουλάχιστον τόσο στο ίδιο ύψος όσο το πάγιο ποσό που πήραν από την Κομισιόν. Δηλαδή έτσι και αλλιώ πρέπει να ε, τηρούνται ε, τα λογιστικά στοιχεία. Άρα δηλαδή τι νόημα έχει αυτό το να ορίζονται ευθύ εξ αρχή εφάπαξ ποσά. Βεβαίω, ε, πρέπει να πούμε ότι το σύστημα αυτό του πραγματικού κόστου ε, είναι διαφανές ε, και βοηθάει στου περισσότερου που συμμετέχουν σε προγράμματα. Θα πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που έχει σχέση με την επιστοποίηση μεθόδου. Εδώ είχε, είχαν υπάρξει πολλές ελπίδες για απλούστευση. Υπάρχουν, όπω ξέρετε, δύο διαδικασίε πιστοποίηση. Η μία όταν χρησιμοποιεί κανεί το μέσο κόστο προσωπικού και η άλλη μέθοδο είναι περισσότερο διευρυμένη, ένα σύστημα εκτεταμένο όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη δική του τη μέθοδο, την οικονομική, που την έχει πιστοποίησει από ε, την Κομισιόν και εκεί υπολογίζει κανείς ε, τις δαπάνες του. Μετά από μια μεγάλη καθυστέρηση 2,5 ετών, επιτέλους η Κομισιόν τον Ιούνιο του 2009 τροποποίησε τα κριτήριά της ε, για να μπορεί να γίνεται χρήση αυτού του μέσου κόστου προσωπικού. Πρέπει όμω να πω ότι μέχρι τώρα οι ενδείξει κατατείνουν στο ότι κανεί δεν καλύπτει ε, τα, ορισμένα, τα καθορισμένα κριτήρια. Ε, και αυτά ίσως ε, είναι καλά στοιχεία για τις μεγάλες εταιρείες. Από εκεί οι εταιρείε μπορούν να πάρουν ε, κάποια χρήσιμα στοιχεία. Ίσως εδώ ε, επιθυμώ να αφαιρθούν οι συνάδελφοί μου από τις μεγάλες βιομηχανίες. Όσον αφορά όμως τις, ε, τους ε, οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας. Εμείς ως Ομοσπονδία πήραμε στοιχεία από 30 μεγάλους οργανισμούς και από εκεί καταλήξαμε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών χρησιμοποιούν αυτό το κόστος όταν χρεώνουν ε, έρευνα και τεχνολογία σε τρίτα μέρη. Το 80% των 30 αυτών μεγάλων οργανισμών κατηγορηματικά δεν μπορούν να καλύψουν τα κριτήρια τα οποία έχει ορίσει η Κομισιόν. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους οργανισμούς δεν νιώθουν ότι μπορούν να καλύψουν τα κριτήρια και δύο από τους 30, έτσι κι πριν από αρκετούς μήνες αποφάσισαν ότι ενώ στο ε, έκτο πρόγραμμα χρησιμοποίησαν αυτό μέσο κόστος, στο έβδομο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουν ε, εξατομικευμένο κόστος προσωπικό και θα σε εξηγήσω γιατί θα το κάνουν αυτό ε, ευθύ αμέσω. Άρα δηλαδή, εάν οι κανόνες για τη μέθοδο περί μέσου κόστους προσωπικού δεν αλλάξουν ριζικά, αυτή είναι μια απλούστευση άχρηστη θα έλεγα, γιατί σχεδόν κανείς δεν μπορεί να καλύψει τα κριτήρια. Και ε, η μέθοδος αυτή ούτε, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά εμποδίζει και στο να υπάρχει ένα μέσο κόστος ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε συγκεκριμένα παραδείγματα απλούστευσης ε, και στο πιστοποιητικό ελέγχου. Εδώ πρέπει να πω έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Γιατί ε, τα πιστοποιητικά που πρέπει να καταβάλουν ε, οι ανάδοχοι στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με το έκτο πρόγραμμα. Και αισθάνομαι όμως ε, ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί βέβαια και αυταπάτη. Και εδώ αναφέρομαι στην εκστρατεία της Κομισιόν για τους ελέγχους του έκτου προγράμματος και για το ότι έχει πει θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι και για το πρόγραμμα 7. Ε, θεωρώ ότι η πρακτική συνέπεια είναι ότι στο μέλλον τα πιστοποιητικά ελέγχου θα είναι σε μεγάλο βαθμό περιτά, γιατί θα έχουμε έτσι κι αλλιώς άμεσο έλεγχο από την Επιτροπή. Φτάνουμε τώρα στη, σιγά σιγά στην ουσία του προβλήματος. Η εκστρατεία περί ελέγχου της Κομισιόν για το 7ο πρόγραμμα διενεργείται με τέτοιο τρόπο που ε, πραγματικά έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή, στρεβλώνει, ε, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη προς την Κομισιόν ως ένα αξιόπιστο εταίρο στην έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζημιώνει τις ε, συνεργασίες, ε, συνεργασίες που σφυριλατήθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια και σε πολλά προγράμματα πλαίσιο, αυξάνει το διοικητικό άχθος και τέλος φαλκιδεύει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθιστώντας τη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο όλο και λιγότερο ελκυστική. Για να είμαι λοιπόν ειλικρινής υπάρχει αυτό το κλίμα της ε, δυσπιστίας ε, που διαμορφώνεται και οι συνέπειες είναι διαβρωτικέ, ε, ιδιαίτερα αρνητικέ. Άρα δηλαδή πρέπει αυτό να σταματήσει επιγόντω, γιατί ε, αλλιώ όλο και λιγότεροι οργανισμοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο 7ο πρόγραμμα. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα της ε, δυσπιστία. Πριν από λίγο ανέφερα δύο οργανισμού έρευνα και τεχνολογία, που αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τα κριτήρια τη Κομισιόν για το μέσο κόστο προσωπικού και εν πάση περιπτώσει αποφάσισαν ότι προτιμούν, παρότι προτιμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το μέσο κόστο προσωπικού στο πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 δεν θα το κάνουν τελικά. Θα χρησιμοποιήσουν εξατομικευμένο κόστο. Και παρότι χρησιμοποιούν, όπω σα είπα, το μέσο κόστο προσωπικού στα εθνικά προγράμματα, ε, και όταν εργάζονται για άλλους τρίτους δεν θα το κάνουν με την Κομισιόν. Ο λόγος είναι γιατί δεν εμπιστεύονται πια την Κομισιόν. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία των ορισμών της Κομισιόν για το ποιο είναι το, ε, το αποδεκτό κόστος. Αυτό που σήμερα μπορεί να είναι αποδεκτό κόστος, μετά από 6 μήνες μπορεί να πάυσει να είναι. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να έχουν μια ελάχιστη νομική ασφάλεια και αυτή η ελάχιστη νομική ασφάλεια δεν είναι πλέον δεδομένη. Για να κατανοήσει λοιπόν κανείς όλα αυτά, πρέπει να κατανοήσει και τη φύση και τις ε, συνέπειες ε, της εκλογικής, της εκστρατείας της ε, Κομισιόν για τους ελέγχους. Η εκστρατεία αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο που de facto η Κομισιόν λειτουργεί αναδρομικά, μόνο μερός αλλάζει τον ορισμό του αποδεκτού κόστους. Κόστος που η ίδια η Κομισιόν κατά το παρελθόν είχε αποδεχθεί. Και θα σα εξηγήσω περί τίνο πρόκειται. Αλλά να είμαστε σαφεί. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που περιορίζεται σε ε, ένα ή δύο μετέχοντε στο έκτο πρόγραμμα. Είναι ένα εκτεταμένο πρόβλημα και θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά παραδείγματα και αριθμού. Από του 20 ε, συμμετέχοντε στο έκτο πρόγραμμα υπάρχουν πολλοί οργανισμοί έρευνα και πολλέ ε, βιομηχανικέ εταιρείε, οι οποίε σύμφωνα με την Κομισιόν και με τι πληροφορίε που έχω προλάβει εγώ και μετά από ελέγχους που έγιναν σε ε, project ε, όπου συμμετείχαν αυτοί οι οργανισμοί και οι εταιρείε ή εξακολουθούν να συμμετέχουν ακόμα, μετά από όλα αυτά ε, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν συστηματικά λάθη στον υπολογισμό του κόστου των δαπανών. Και για πολλά χρόνια κάθε ένα από αυτού του οργανισμού, το κόστο τη δαπάνε, τις ανέφεραν στην Κομισιόν χρησιμοποιώντα συστηματικά του ίδιου ορισμού, την ίδια μέθοδο για να γίνει ο υπολογισμό του κόστου με άλλα λόγια, ε, στην γλώσσα τη δική μας ε, λειτουργήσαν σωστά, αποδεκτά με βάση τα κριτήρια της λογιστικής. Μετά όμως από τους ελέγχους η Κομισιόν λέει ότι οι ε, αποδέκτες έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη και τους ζήτησαν να ξανακάνουν τους υπολογισμούς των δαπανών για όλα τα προγράμματα. Και εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο εργασία. Ε, κατά κανόνα χρειάζεται κανεί 45 μέρε για να το κάνει αυτό και το λογαριασμό τον πληρώνει μόνο του. Και ένα από τα μέλη μα πλήρωσε 75.000 ευρώ για να προσλάβει μια ομάδα ορκωτών λογιστών από την από την γνωστή αυτή εταιρεία ελεκτών ορκωτών λογιστών που θα κάνει τους ελέγχους. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτούς τους αριθμούς και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Λίγες είναι περιπτώσεις εκείνες ε, από τους ε, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που είναι ικανοποιημένοι. Αυτά λοιπόν όλα αφορούν συμμετοχές, περίπου 2.700 συμμετοχές. Κάθε πρόγραμμα ε, περιλαμβάνει τρία στοιχεία δαπανών. Έχουμε 7.500 στοιχεία κόστους που ε, έχει γίνει αποδεκτό από την Κομισιόν και έχει υπογραφεί από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους ε, της ε, Κομισιόν, των ε, Project και των Financial Officer. Έχουμε λοιπόν χιλιάδες υπογραφών από πλευράς Κομισιόν. Είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για έναν ή δύο υπαλλήλους Κομισιόν που ενδέχεται να έκανε κάποιο λάθος στο να υπογράψουν, να προσυπογράψουν την διασταύρωση των στοιχείων που υποτίθεται είχαν λάθη. Όχι, μιλάμε για εκατοντάδες υπαλλήλων της Κομισιόν. Και το μόνο συμπέρασμα που μπορεί κανείς να εξάγει από όλα αυτά είναι ότι η Κομισιόν ε, τελικά απέτυχε ε, στο να υπολογίσει τις δαπάνες του έκτου προγράμματος. Ε, μιλάμε για ανάδοχους που λειτουργήσαν με καλή πίστη και η Κομισιόν Βεβαίω και αποδέχθηκε επανειλημμένα τη δική του συμπεριφορά προ υπογράφοντα ε, τι δαπάνε. Αν έγιναν λάθη, έγιναν λάθη και από την Κομισιόν. Τώρα όμω φαίνεται η Κομισιόν θεωρεί ότι μόνο οι ανάδοχοι, οι εμπλεκόμενοι θα πληρώσουν τα δικά, πληρώσουν τα δικά τους λάθη. Αυτή είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Και όπω σα είπα προηγουμένω, η Κομισιόν αναδρομικά και μονομερός αλλάζει τον ορισμό του αποδεκτού κόστους. Από νομικής πλευράς τέτοιου είδους συμπεριφορά αντιβαίνει με βασικές αρχές ε, του δικαίου περί συμβάσεων και Ίσως για πρώτη φορά να ακούτε ότι δύο από τους ερευνητικούς οργανισμούς στους οποίους αναφέρθηκα αποφάσισαν να καταφύγουν ε, στο δικαστήριο και να ενάγουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι λοιπόν, ε, από πού προκύπτει το πρόβλημα και τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρόβλημα προκύπτει για διάφορους λόγους. Το θέμα είναι ότι οι κανονισμοί περί συμμετοχής δεν ε, ορίζουν λεπτομερώς την, το αποδεκτό κόστος αναφέρουν μόνο τις ε, βασικές αρχές, ότι το κόστος πρέπει να είναι πραγματικό, να είναι οικονομικό, ε, να είναι απαραίτητο και να ε, συμβαδίζει με τα βασικά στοιχεία και βασικές αρχές περί λογιστικής. Πολλά δικαστήρια έχουν επικρίνει αυτούς τους ασαφείς κανονισμούς ή Κομισιόν φαίνεται ότι είναι υποπίεση να χρησιμοποιεί και αυτή σαφείς ορισμούς. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτό που κάνει ο νομοθέτης ε, είναι ότι στο παρελθόν υπολόγιζε πάντα την στάση της Κομισιόν όταν καθόριζε το κόστος και για να ερμηνεύσει κανείς αυτές τις ε, γενικές αρχές αναγκαστικά έπρεπε να υπάρχει ε, ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Η Κομισιόν πρέπει να έχει κατά νου τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, στα είδη των οργανισμών. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι τώρα πλέον δεν επιτρέπει επιτρέπεται αυτό, η μία πλευρά θα πρέπει να καλύπτει πάντα, αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό. Άρα δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να προτείνω να διαχωρίσουμε το παρελθόν από το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν αφορά το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και εδώ στην ψηφορία απαλλαγής ε, του προπολογισμού του 2008 σύστησε στην Κομισιόν ως ε, ε, εργαλείο για ε, νομική ασφάλεια να μην ξαναγίνουν νέοι ορισμοί για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο που έχει ήδη ε, τακτοποιηθεί. Αυτή ήταν μια πολύ σαφής σύσταση. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να κάνουμε τους ελέγχους όπως γίνονται τώρα, θα βλάψουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή έρευνα ε, από ότι θα ωφελήσουμε τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έγιναν λάθη στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, έγιναν από όλες τις πλευρές και έγιναν με καλή την πίστη. Αυτό λοιπόν το γεγονός πρέπει να το αποδεχθούμε. Ας πάψουμε να προσπαθούμε να διορθώσουμε το παρελθόν, α τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και ας δούμε το μέλλον. Το μέλλον είναι το επόμενο πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με σωστούς ορισμούς. Και αυτό είναι χρονοβόρο. Επειδή λοιπόν είναι χρονοβόρο, γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι ο στόχος είναι το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ίσως να πρέπει να ε, εκπονήσουμε έναν καινούργιο οικονομικό κανονισμό για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εκείνο που σίγουρα χρειαζόμαστε είναι σαφέστερους ε, κανονισμούς ε, για τη συμμετοχή. Και χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ελέγχων που θα αναγνωρίζει ότι η έρευνα δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως το να επιδοτεί κανείς ε, ε, την κτηνοτροφία ή να συμμετέχει σε δημόσια έργα. Πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω, αν μου επιτρέπετε, οι ευρωβουλευτές και πιο συγκεκριμένα οι, τα μέλη αυτής της Επιτροπής και κυρίως της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών να αναλάβουν την πρωτοβουλία να καλέσουν Υπάρχουν εδώ ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλοι από κοινού να συζητήσουν και να ορίσουν και να συμφωνήσουν για μια ελάχιστη διαχείριση και ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο ελέγχου για τα ερευνητικά προγράμματα. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι ε, των άμεσα ενδιαφερόμενων οργανισμών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα συμπεράσματα αυτής της δουλειάς θα έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ε, το να υψώνει κανεί ε, το δάχτυλο τη ε, κατηγορία και να λέει αυτός ο α ή ο β αυτό έχει περάσει. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Φτάνουμε λοιπόν στο παρόν. Το παρόν είναι το έβδομο πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, οι ανάδοχοι χρειάζονται μια ελάχιστη νομική ασφάλεια. Κάποιο είπε κάποια μέρα η απλούστευση πάνω απ' όλα ε, πρέπει να έχει άμεση σχέση με τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα. Αν τελικά συμφωνήσουμε όλοι να δουλέψουμε για ένα καλό πλαίσιο για το 8ο πρόγραμμα, αυτό που εντωμεταξύ χρειαζόμαστε είναι μια ανοχή, ανεκτική συμπεριφορά και ρεαλιστική προσέγγιση προ το 7ο πρόγραμμα. Αν όλε οι πλευρέ έχουν καλή θέληση, αυτό δεν θα είναι δύσκολο. Υπάρχει η βάση στου κανόνε ε, τη ε, συμμετοχή στο άρθρο 31.3c, 3γ, όπου αναφέρεται ότι αποδεκτό το κόστος είναι εκείνο που ορίζεται με βάση τα την πεπατημένη στη λογιστική ε, και σε αυτά που χρησιμοποιεί ο μετέχων ο ενδιαφερόμενος. Θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να συμβάλλετε και εσείς στο να προοδεύσει η έρευνα, γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο επήγει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που μας είπατε. Θα ήθελα να σας πω τώρα η διερμηνία η στη γερμανική γλώσσα περνάει από την καμπίνα παριθμών 7. Όποιος θέλει να ακούσει γερμανικά παρακαλώ το κανάλι 17. Μετά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Λας Πάλεσεν, πρόεδρο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας. Σας παρακαλώ να τηρήσουμε το χρόνο που έχει ο καθένα στη διάθεσή του, 10 με 15 λεπτά, γιατί αλλιώ ακόμα το απόγευμα εδώ θα είμαστε. 10 με 15 λεπτά παρακαλώ, αλλιώς οι συνάδελφοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Κύριε Πάρεσεν, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορώ σήμερα να σας απευθύνω τον λόγο. Εγώ δεν εκπροσωπώ μια ένωση πανεπιστημίων. Εκπροσωπώ μόνο το πανεπιστήμιο μου, το πώς το βλέπουμε εμείς. Νομίζω όμως πως οι απόψεις μου λίγο πολύ ανταποκρίνονται στο πώς τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνία μάλλον της Ευρώπης βλέπουν αυτά τα ζητήματα. Αυτό το οποίο βλέπετε εκεί κάτω δεξιά δεν είναι το πώς φαντάζεται ένας καλλιτέχνης στη γραφειοκρατία, είναι απλά έτσι λίγη, μια εικονογράφηση από το πανεπιστήμιο μας. Λοιπόν, είναι πολύ λίγα πράγματα για το πανεπιστήμιο μου. Ιδρύθηκε το 1829 από τον φυσικό και χημικό Hans Christian που περιέγραψε τον ηλεκτρομαγνητισμό, ήταν λόγιος και Ευρωπαίος και για την εποχή του δημοσίευσε το έργο του στα δανέζικα, αλλά το περισσότερο στα αγγλικά, αγγλικά και γερμανικά, το μεγαλύτερο όγκο του έργου του και ήξερε και άλλες γλώσσες. Ήταν ένας πραγματικός Ευρωπαίος και εμείς ε, θεωρούμε πως είμαστε οπωσδήποτε ένα διεθνές πανεπιστήμιο που βρίσκεται βεβαίως στη Δανία αλλά έχει διεθνή εμβέλεια. Έχουμε γύρω στους 6.500 φοιτητές, ε, λίγο περίπου όσο το MIT και άλλα πολυτεχνία να έχουμε προσωπικό 4.500 άτομα, 2.500 από τα οποία είναι ερευνητές και άλλους χίλιους υποψήφιους διδάκτορες. Χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω, θα έλεγα ότι είμαστε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο με διεθνές προφίλ. Ο δε ο δε δείκτης του Λάιντεν που βασίζεται μόνο στην έρευνα μας έχει κατατάξει τα πέντε πρώτα πανεπιστήμια της ε, Ευρώπης. Το πέμπτο για την ακρίβεια μεταξύ των 100 μεγαλύτερων. Επίσης είμαστε ο μεγαλύτερος δικαιούχος στην Δανία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με 29 εκατομμύρια ευρώ το 2008. Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από πλευράς οικονομίας, οικονομιών. Ε, εγώ τώρα, βεβαίως δεν θα αναφέρω μόνο τα λάθος τι λάθος ε, πτυχές θεωρούμε πως οι περισσότερες πτυχές του προγράμματος πλαισίου 7 είναι εξαιρετικέ η χρηματοδότηση είναι εξαιρετική, η ιδέα του να υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια είναι θαυμάσια. Οπότε θα δεχτούμε και τη γραφειοκρατία. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό το να ενώσει η Ευρώπη τις ε, δυνάμεις της. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, όλες οι εφευρέσεις που θα εμπλουτίσουν την ανθρωπότητα θα γίνουν στην Άπο Ανατολή ή στη ΣΥΠΑ. Έχω καλούς φίλους ε, και στην Άπο Ανατολή και στις ΙΠΑ. Ε, Οπότε βεβαίω και αυτοί θέλουν να προωθεύσουν οι περιοχές τους, αλλά εάν εμείς δεν κάνουμε κάτι ως Ευρωπαίοι, και νομίζω ότι κάνουμε, θα μείνουμε πίσω. Δεν είναι γραμμένο ότι δεν μπορούμε εμείς σε 30 ή 40 χρόνια να μην είμαστε η φτωχότερη περιοχή του πλανήτη. Όχι σε 100, σε 30-40 χρόνια μπορούμε να είμαστε η φτωχότερη περιοχή του πλανήτη. Αυτό δεν θα συμβεί εάν συνεχίσουμε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο, λόγο, ρόλο με που έχουμε. Και πριν περάσω στις βελτιώσεις που θα ήθελα εγώ να τονίσω πως το πρόγραμμα πλαίσιο 7 είναι μεγάλη επιτυχία και το εκτιμούν πάρα πολύ τα πανεπιστήμια. Τώρα, να περάσω στα σημεία εκείνα τα οποία χρειάζονται βελτίωση. Το πρόγραμμα πλαίσιο 7 μέχρι στιγμή έχει 160.000 συμμετέχοντες που έχουν ζητήσει χρηματοδότηση και 35.000 βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σύμβασης. Εάν κάνουμε μικρές μόνο βελτιώσεις, έτσι ώστε ο κάθε ένας από αυτούς να γλιτώσει δύο μέρες διοικητικής εργασίας, τότε αυτό ανταποκρίνεται σε 2.240 ανθρωποέτη. Δηλαδή όσο είναι η ετήσια ε, ποσότητα ας της έρευνας στο πανεπιστήμιό μου. Οπότε κλειδώνουμε κάτι. Και είναι εύκολο να γίνει αυτό. Να περάσω τώρα σε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Δεν πρέπει μόνο να γλιτώσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, πρέπει να αυξήσουμε και την ποιότητα. Και εμείς θεωρούμε πως ε, πολλές από τις εκκλήσεις και πολλές από τις προκηρύξεις είναι πολύ περιορισμένες. Και συνήθως ε, εννοείται πως θα χρηματοδοτηθεί μόνο μία πρόταση. Είναι γνωστό ε, αυτό στους ερευνητές. Ε, και όταν ξέρουν πως ε, θα χρηματοδοτηθεί μόνο μία πρόταση ανεξαρτήτως του ότι μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις ε, πολλά υποσχόμενες προτάσεις μπορούν να πούν δεν θα ασχοληθούμε γιατί ξέρουν πως υπάρχουν δύο-τρεις άλλοι συνάδελφοι που θα καταθέσουν αίτηση οπότε τι συμβαίνει έχουμε λιγότερες ποιοτικέ αιτήσει. αυτό είναι κρίμα πολλοί από τους καλύτερους ερευνητές δεν υποβάλλουν όσες προτάσεις θα μπορούσαν, αλλά ασχολούνται με έναν τομέα μόνο και αν δεν πάρουν εκεί τη χρηματοδότηση θα απογοητευτούν και θα στραφούν σε εθνικές πηγές. Που, εντάξει, θετικό μπορεί να είναι αυτό, αλλά δεν είναι το σκεπτικό εδώ το ευρωπαϊκό. Η σύστασή μας είναι να ορίσουμε ευρύτερα θέματα με τον ανάλογο προϋπολογισμό για να μπορούν να χρηματοδοτηθεί πέραν του ενός έργου σε κάθε τομέα. Επίσης κάτι άλλο που είναι εύκολο νομίζω να γίνει είναι οι προκηρύξεις να μην δημοσιεύονται ταυτόχρονα και οι προθεσμίες να είναι εντός δύο μηνών. Ε, δείτε το πρακτικά. Η γραμματεία σε κάθε πανεπιστήμιο θα πιεστεί πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο μήνους και πρέπει εμείς να τους προσλάβουμε και τους πληρώνουμε για ένα ολόκληρο χρόνο. Δεν χρησιμοποιούμε έτσι αποτελεσματικά τα κονδύλια. Ξεκολώνονται, με συγχωρείτε. Ε, θα πρέπει να δουλεύονται ολόκληρο το χρόνο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται και στο δικό μου πανεπιστήμιο και στα υπόλοιπα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και είναι κάτι που επίσης είναι εύκολο να γίνει. Κατόπιν. Εναρμόνιση κανόνων και διαδικασιών. Έχουμε διαφορετικούς ε, κανόνες και διαδικασίες για κάθε πρόγραμμα, για τις ε, κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίε, για την έρευνα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλοι κανόνες. Συνεργασία, πάλι άλλοι κανόνες. Είναι αντιπαραγωγικό, γιατί κατά την εμπειρία μου μετά διαλέγει ο καθένας. Εντάξει, καλό είναι να διαλέγει κανεί όταν μπαίνει σε ένα ε, φούρνο, αλλά ε, αντιλαμβάνεστε, δεν έχει άλλα χρήματα για το φούρνο και άλλα για το χασάπικο κτλ. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν το ότι παντού ισχύουν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα, περνάει το ίδιο νόμισμα. Οπότε οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί και να μην διαλέγει κανείς εκεί που είναι ευκολότεροι οι κανόνε να υποβάλει αίτηση. Και νομίζω ότι από αυτό υποφέρει το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξενορίζω πως είναι περίεργο αυτό το σχόλιο από μια χώρα που δεν έχει ακόμα υιοθετήσει το ευρωπαϊκό νόμισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τόσο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα άλλο ελάττωμα για την έρευνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πως δεν είναι πολύ ισορροπημένοι οι όροι. Δηλαδή για να διασφαλιστούν οι κανόνες αυτοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολοι οι κανόνες εις βάρος των πανεπιστημίων και της έρευνα. Γιατί εμποδίζεται η ελευθερία δράσης. Οι κανόνες είναι τέτοιοι ώστε πάρα πολλά πανεπιστήμια έπρεπε να μεταφέρουν τα δικαιώματα Πνευματική ιδιοκτησία σε κάποιον άλλον και δεν θα μπορούσαν να κάνουν έρευνα σε αυτόν τον τομέα στο μέλλον. Κανένα πανεπιστήμιο δεν θα δεσμεύονταν ότι δεν θα ερευνήσει αυτόν τον τομέα πλέον στο μέλλον. Ξέρω πώ αυτό γίνεται για να ωφεληθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Αλλά τα πανεπιστήμια δεν θα ασχοληθούν με αυτόν τον κανόνα, με τον να ε, δίνεται λοιπόν αυτή την ευνοϊκότερη μεταχείριση μικρομεσαίε επιχειρήσει, δεν θα ασχοληθεί κανεί μαζί του. Επίση, θεωρούμε πως ε, καλό θα ήταν το περιθώριο ερμηνείας που έχουν είχε οι στην Κομισιόν θα πρέπει να περιοριστεί. Εμείς θεωρούμε πως είναι πολύ προσωπική και υποκειμενική η εφαρμογή των κανόνων. Δηλαδή αν αλλάξει ο αρμόδιος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι προφανές πως είναι υποκειμενική η διαδικασία. Και αυτό δεν είναι λογικό και δεν είναι πρακτικό γιατί στέλνει ένα μήνυμα αβεβαιότητας στην ερευνητική κοινότητα. Έχω κατόπιν άλλη μια πρόταση και γνωρίζω πως όσοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα θα πούνε πως είναι γελίο αυτό και δεν έκανα όλη αυτή την, την εισαγωγή για να, πει, για να μην πει κάποιος ότι δεν είναι γελίο γιατί ξέρω πως θα το πούνε στη δική σταδιοδρομία μου έχω περάσει από διάφορες θέσεις, από τη βιομηχανία, το πανεπιστήμιο, σε κάτι ενδιάμεσο και συχνά βρίσκομαι σε οργανισμούς όπου η άποψη του οργανισμού είναι πως λειτουργεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Και όταν ήρθα εγώ ως νέος διευθυντής και είπα θα τα αλλάξουμε αυτό, λέγανε πάντα «Α, όχι, αυτό δεν γίνεται, το έχουμε ξαναδοκιμάσει και δεν γίνεται. Και εκεί πέρα χρειάζεται ένα ηγετικό ρόλο. Η εμπειρία μου δείχνει πως σε κάθε οργανισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξοικονομηθεί ένα 5%. Είναι αδύνατο να εξοικονομηθεί ένα 2%, αλλά 50% είναι πολύ εύκολο. Το 2% είναι αδύνατο γιατί μπαίνουμε σε πολύ ψηλό πράγματα. Δηλαδή ε, χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μολύβια, γράφουμε και στην πίσω μεριά των σελίδων και μετά από λίγο δεν επιτυγχάνεται ούτε το 2%. Το 5% είναι κάπως ευκολότερο γιατί πρέπει να σκεφτούμε. Αλλά το 50% είναι πανεύκολο. Γιατί πρέπει να ξανασχεδιαστεί το σύστημα από την αρχή. Οπότε εκεί χρειάζεται δημιουργικότητα και οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί όταν χρειάζεται. Έχω λοιπόν κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν αφελείς και μπορεί να θεωρείτε πως απλά δεν ξέρω το τι γίνεται, αλλά θα τα προτείνω παρόλα αυτά. Πρώτη σύσταση, να είναι σταθερή η προθεσμία 60 ημέρες για την αξιολόγηση των νητήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100, γύρω στις 129 μέρες. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό με το να βρίσκουμε γρηγορότερα τους ε, αξιολογητές, αλλά για να μείνω στην εμπειρία του παρελθόντος, ως οι κορυφαίοι εσείς ενός οργανισμού δεν πρέπει να προτείνετε λύση, πρέπει να ζητήσετε αυτό το αποτέλεσμα ότι θέλετε. Να πείτε 60 ημέρες, να το μειώσουμε στα δύο και όταν έρθουν οι γραφειοκράτες και σας πούνε είναι αδύνατον, τότε να τους πείτε ξαναπροσπαθήστε. Και αν ξανάρθουν και σας πούν δεν γίνεται, τότε ως πολιτικοί πρέπει να πείτε «Ε, πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τότε να κάνουν τη δουλειά μας. Έτσι κάνουμε στις επιχειρήσεις και στο πανεπιστήμιο. Δεύτερη σύσταση. Να υπάρχει σταθερή προθεσμία 60 ημερών για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση. Τώρα είναι 200 ημέρες. Είναι πάρα πολύ. Και πάλι η εμπειρία μου λέει πως ε, συχνά ο περισσότερος χρόνος δεν σημαίνει καλύτερη ποιότητα. Έτσι, και λίγη βιασύνη χρειάζεται. Ε, το να υδρώσει κάποιος λίγο ωφελεί. και πάλι μπορείτε να πείτε πως ε, μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες οι χειριστές δύο φορές μόνο. Οπότε εκεί πέρα θα σκεφτούν πάρα πολύ καλά το τι θα ρωτήσουν την πρώτη φορά και πολύ περισσότερο τη δεύτερη που θα είναι η τελευταία φορά που θα ζητήσουν πληροφορίες. Και όταν τους δοθούν οι περαιτέρω πληροφορίες θα τους πείτε έχετε 10 μέρες. Θα σου πούν δεν μπορούμε, θα λυπούμε μετά, η αίτησή σας απορρίπτεται. Σας υπόσχομαι τα πανεπιστήμια σε 10 μέρες θα απαντήσουν. Το δικό μου το πανεπιστήμιο, ακόμα και αν χρειαστεί να δουλέψουμε Σαββατοκύριακα. Και όταν τελειώσει θα είμαστε ικανοποιημένοι γιατί θα έχουμε μια θετική απάντηση σε λιγότερες ημέρες αντί για 129. Ναι ή όχι. Νομίζω ναι, εν πάση περιπτώσει. Κατόπιν για μικρότερα ερευνητικά ιδρύματα από το πανεπιστήμιό μου, καλύτερο θα ήταν να αυξηθεί η διαφάνεια μέσω ενός εγχειριδίου, το οποίο θα περιέχει τις διαπραγματεύσεις, τις συμβατικές, με κάποια ορόσημα, με κάποια σταθερά σημεία, για να παρακολουθούν τη διαδικασία. Σε μεγάλες εταιρείε, σε μεγάλους οργανισμούς, αρέσει η γραφειοκρατία. Γιατί, Γιατί έτσι αποκλείονται οι μικροί ανταγωνιστές. Ε, δεν θέλουμε όμως αυτό στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουν όλοι. Οπότε πρέπει να είναι εύκολο και για τους μικρότερους οργανισμούς που δεν έχουν εμπειρία. Νομίζω αυτό μπορεί να βοηθήσει εκεί. Κατόπιν. Εντάξει, εγώ προέρχομαι και από πολυτεχνείο, το φαντάζεστε, βλέπετε εδώ πέρα, να αναπτυχθεί και να υπάρξει ένα σύστημα online για την κατάθεση προσφορών, τη διαπραγμάτευση και τις, ε, την παρακολούθηση. Εύκολο αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από το πρόγραμμα ε, ICT, τεχνολογίας ε, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, και ο κύριος Χαλ το ίδιο ανέφερε, να περάσουμε από το 60% στο μοντέλο του πλήρους κόστους. Σε αυτό θα πρέπει να μείνουμε. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα γιατί δεν γίνεται. Δε, Πλήρες κόστος. Είναι καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύτερο για τους λογιστές το ευκολότερο και να θυμάστε πως η έρευνα διαφέρει πάρα πολύ από τις επιδοτήσεις στη Γεωργία ή κάπου αλλού. Να θυμάστε πως αυτό το οποίο πρέπει να ελέγχεται και είναι σημαντική η έλεγχη είναι το αποτέλεσμα της έρευνας. Τώρα ελέγχεται το εάν ε, μπορούμε να φέρουμε απόδειξη για το εάν πήραμε λεωφορείο ή ταξί. Δεν λέω πως δεν είναι σημαντικό, αλλά περίπου αυτό λέω. Δεν είναι πιο σημαντικό να υπάρχουν κάποιοι επιστημονικοί ας πούμε λογιστές να πούνε τι αγοράζουμε με αυτά τα λεφτά, έχουμε έρευνα και τα υπόλοιπα μετά η μικροδιαχείριση να μείνουν στο ελάχιστο. Αλλά να ελέγχεται το ότι πραγματικά υπάρχει έρευνα ως αποτέλεσμα. Αυτό θα θέλαμε εμείς και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που τηρήσατε ακριβώ το χρόνο σα. Ο επόμενο εκπρόσωπο βιομηχανία, Γιάνν Φανεμπίζεν, έρευνα και τεχνολογική καινοτομία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 Σα Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Έκα, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσω ευχαριστώντα τα μέλη της Επιτροπής ΕΤΡΕ που κάλεσε την Business Europe να σα μιλήσει εδώ. Η Business Europe εκπροσωπεί πάνω από 20 εκατομμύρια μικρέ και μεγάλε επιχειρήσει στην Ευρώπη. Ας αναφέρουμε πρώτα τα θετικά. Πιστεύουμε ότι πολλές εταιρείες μπορούν και πραγματικά ωφελούνται με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα. Ε, μια από τις κύριες ισχύες ε, των προγραμμάτων είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας με εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Μειώνεται δηλαδή ο κίνδυνος τα δημόσια χρήματα δίνουν στην δυνατότητα στις εταιρείε να κάνουν περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη από ό,τι θα μπορούσαν κανονικά. Η συμμετοχή ενθαρρύνει στην δημιουργία και εφαρμογή νέων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και πρόσβασης σε προηγμένα ερευνητικά κέντρα και υποδομές. Η συμμετοχή αυτή ενθαρρύνει την κοινοτικότητα των επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ των εταιριών και των ερευνητικών Ινστιτούτων. Και κάτι επίσης σημαντικό είναι το πρόγραμμα πλαίσιο ε, δίνει ένα ε, πιστό περιβάλλον, προσφέρει ένα πιστό περιβάλλον, πράγμα που είναι σημαντικό σήμερα που υπάρχει αυξημένη συνεργασία που αποτελείται ανοιχτή καινοτομία. Οποιοδήποτε ερευνητή στην Ευρώπη μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε άλλο συνάδελφό του για να συνεργαστούν. Και η συνεργασία που απορρέει από αυτό είναι ένα όφελος για την Ευρώπη. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ανέπτυξε κάποια νέα μέσα που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία. Παραδείγματο χάρη ε, το να μοιράζονται το κίνδυνο, οι τεχνολογικές, οι κοινές ε, ε, πρωτοβουλίε που είχαν ξεκινήσει μέσα στα πλαίσια του έκτου προγράμματο ήδη. Παρ' όλα αυτά, παρόλο το δυναμικό αυτό για όφελος, η συμμετοχή τη βιομηχανία μειώνεται τα 15 τελευταία χρόνια. Η μείωση ξεκίνησε από 39% στο τέταρτο πρόγραμμα σε 31% στο πρόγραμμα 6 και για το πρόγραμμα 7 αυτή τη στιγμή η συμμετοχή είναι της τάξης του 25%. Προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί ε, έγινε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία στη συμμετοχή των ε, επιχειρήσεων. Τρει συγκεκριμένοι τομεί ανησυχία για τι εταιρείε. Οι κανόνε είναι πολύπλοκοι και χρονοβόροι για τη συμμετοχή. Το θέμα του μέσου κόστου για το προσωπικό και κατά τρίτον υπερβολική γραφειοκρατία. Όπω φαίνεται και στην περίπτωση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Κάθε ένα από του τομεί αυτή είναι αντίθετος από τις προσπάθειες της ε, επιχειρησιακή κοινότητα, όπου η αύξηση της αποτελεσματικότητα αποκτά όσο πάει και μεγαλύτερη σημασία εν ώψη του διεθνούς ανταγωνισμού. Είναι πολύπλοκα τα θέματα, ο κίνδυνος δεν είναι αρκετά επαρκής, και εμείς προσπαθήσαμε πολλά για να απλουστεύσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο παριθμών 7. Φοβόμαστε όμως ότι δεν επιτεύχθη ε, η επιτυχία που ελπίζαμε. Θα αναφερθώ σε σύντομα. <clears throat> Καταρχήν όσον αφορά τους πολύπλοκους και χρονοβόρους κανόνες, υπήρχε κάποια πρόοδος μεταξύ του 6ου και του 7ου προγράμματος. Παραδείγματος χάρη, οι εγγύσεις για την διαχείριση του κινδύνου και η μοναδική δυνατότητα καταγραφής ούτως ώστε οι πληροφορίες που χρειάζονται να χορηγούνται μόνο μία φορά. Παρ' όλα αυτά, η πρόσβαση στο 7ο πρόγραμμα δράσης εξακολουθεί να είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη. Παραδείγματο χάρη, οι κανόνε συμμετοχή είναι πολύ πολύπλοκοι. Υπάρχει περιοδικό αριθμό μέσων, ανισορροπία μεταξύ του αριθμού ακαδημαϊκού και ε, επιχειρησιακού προσωπικού για την αξιολόγηση, όπω είπε και ο σας, έλλειψη εναρμόνιση για την εφαρμογή των κανόνων και των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που οδήγησε σε σύγχυση και η ε, τυχαία ερμηνεία της ε, εντολής που θα πρέπει να δοθεί στους αρμοδίους κάθε σχεδίου. Μετά, το θέμα του μέσου προσωπικού κόστου, κόστους προσωπικού, όπως είπε και ο συνάδελφος. Αυτό είναι ένα θέμα που τώρα όσο πάει και διαφαίνεται και γίνεται όσο πάει και μεγαλύτερη ανησυχία και για τους υπηρεσιακούς τομεί. Μια που οι εταιρείε όσο πάει δρούν διεθνώ, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες που ακολουθούνται ε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες λογιστικών βιβλίων. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος δράσης, ζητούν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία για την κράτηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρεία. Και ανησυχούμε ιδιαίτερα από αυτό που ακούμε ότι η ο Κομισιόν δεν θα δέχεται πια μεθοδολογίες του τύπου cost center ή παρόμοιους μέσους ε, όρους που χρησιμοποιούνται και ε, στι επιχειρήσεις και στα ερευνητικά κέντρα. τα νέα, οι νέες διατάξεις στο πρόγραμμα 7 οδηγεί σε αύξηση του γραφειοκρατικού άχθους. Το κόστος αυτό φτάνει ίσως στα 500.000 ανά έτος και ανά επιχείρηση. Αυτό βέβαια αποτρέπει από τη συμμετοχή. Λυπούμεθα γι' αυτό τη, για την απόφαση της Κομισιόν για το μέσο κόστος που ελήφθη στις 23 Ιουνίου 2009 γιατί δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις παραγράφους 117 και 118 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου τρέχοντος έτος. Και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση σχέση με το έκτο πρόγραμμα δράσης. Τρίτος τομέας η υπερβολική γραφειοκρατία, για παράδειγμα η εμπειρία στην ε, κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Τα ίδια προβλήματα πολυπλοκότητας και γραφειοκρατίας που αναφέρθηκαν για το πρόγραμμα πλαίσιο και μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια πορίσματα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θέλουν το πρόγραμμα πλαίσιο να είναι επιτυχές. Παρ' όλα αυτά η προσέγγιση θα πρέπει να βελτιωθεί πριν ξεκινήσουν νέες κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Ο ε, κύριος Δουτριά θα αναφερθεί συγκεκριμένα στο κοινή, στην κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία Clean Sky. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα άλλο σχέδιο και τα σχέδιά μου αφορούν και την ΕΝΙΑΚ, ένα άλλο τομέα ε, που ασχολείται με άλλα θέματα και όχι ηλεκτρονικά. Κάθε μια από αυτές τις ε, συνεργασίας αφορά κράτη, 20 κράτη-μέλη, την Κομισιόν και ενδιαφερόμενα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Μέχρι στιγμής βασίζεται στο άρθρο 171 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το άρθρο ποτέ δεν είχε ε, χρησιμοποιηθεί για ε, ε, συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η διαδικασία κόστισε πάνω από τρία χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος ενός κοινοτικού φορέα. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το προσωπικό και αυτό οδήγησε σε πολύ βεβαρημένη διαδικασία και σημαντικότητες καθυστερήσεις μέχρι να είναι λειτουργικό το σύστημα. Επίσης, ε, ε, ερευνητές και ε, επιστήμονες που συμμετάσχουν στο σύστημα αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο πολλαπλών εποπτιών και ερευνών μέχρι πάνω από 20. Συστάσεις λοιπόν είναι ότι χρειάζεται απλούσταση των κανόνων και διακασιών όχι μόνο για τα GTI αλλά και για όλο το πρόγραμμα πλαίσιο. Να προσδοθεί η τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που χρειάζονται για συμμετοχή στα σχέδια. Να μειωθεί ο αριθμός και το μέγεθος των επισήμων εγγράφων. Να μειωθεί ο χρόνος για τις πληρωμές μετά που θα υποβληθούν οι εκθέσεις για τα σχέδια Ιδίω για τις ε, ΜΜΕ, όπου να περιμένουν πάνω από τρει μήνες είναι υπερβολικό για να μπορέσουν να πληρωθούν, να εξασφαλιστεί ε, μια ακριβή προτεραιότητα για κάθε ένα θέμα, με κατανομή στο ετήσιο προπολογισμό και να επανεισεχθούν οι ξεχωριστές κατηγορίες που υπήρχαν στο πρόγραμμα πλαίσιο υπερθυμών 5 για τους συνδεδεμένους εταίρους. Θα θέλαμε επίσης η αρχή της υπεύθυνη ε, συμμετοχή να ε, δριωθεί μέσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Τον Οκτώβριο μοιράστηκε ένα εγχειρίδιο σχετικό για το πώς μπορούν αυτά τα συνεργατικά προγράμματα να λειτουργήσουν σωστά. Δεύτερη σύσταση σχετικά με το μέσο κόστος για το πλαθωτικό πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση όσον αφορά το, την, προσωπική, την προσωρινή συγγνώμη, αποδοχή του μέσου όρου αναώρα για το κόστος ανά κέντρο. Ταυτόχρονα η Κομισιόν θα πρέπει να αναθεωρήσει τους ε, οικονομικούς κανόνες του προγράμματος 7 σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 23 ε, Απριλίου 2009 παράγραφοι 117 και 118. Τα μέλη της Επιτροπής του Μεσονομικού Ελέγχου έχουν επαναλάβει πολλές φορές τις ανησυχίες αυτού του κοινοβουλίου στην γνωμοδότησή τους της 1ης Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό όμως, η Business Europe καλεί να υπάρχει μια προσέγγιση που να ανέχεται το κίνδυνο και να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Να μην ξεχνάνε, πάντα η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή όμως το θεσμικό σύστημα που ισχύει υπόκειται κυρώσει από την πολιτική αναγκαιότητα να αποφευχθεί ο κίνδυνος και όχι να ε, προωθηθεί. το κόστος του ελέγχου ξεπερνά τα ωφέλη. Και υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτό το κόστος θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο όταν οι ε, διοικητικές αρμοδιότητες της Κομισιόν για το πρόγραμμα πλαίσιο θα περάσουν στα χέρια τσιτή και άλλων. Οι κύριοι περιορισμοί που παρεμποδίζουν την απλούστευση είναι στον δημοσιομικό κανονισμό. Παραδείγματος χάρη ο μηδενικός κίνδυνος που προωθείται αυτή τη στιγμή προέρχεται ίσως από τις ε, διατάξεις για την προσωπική και οικονομική ευθύνη του προσωπικού. Γι' αυτό μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού οικονομισμού η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πετύχει τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια μάλιστα των περιορισμών αυτών δεν μπορούν να πτύχουν πάνω από το 2% αυτών των μικρών ε, προόδων στην οποία αφέρθηκε και ο προλήσας. Χρειαζόμαστε όμως ένα 50% πρόοδο με μια νέα διατύπωση του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί ο δημοσιονομικός κανονισμός και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προβλεπόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για να δημιουργηθεί μερική εξέλιξη για την έρευνα και την καινοτομία για να προβλεφθεί αποδοχή ενός κινδύνου που οπωσδήποτε ελοχεύει καθημερινά στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Επίσης, ε, δεν υπάρχει στο κίνδυνο καθόλου η ιδέα του ιδιωτικού εταίρου που θα πρέπει όμως να υπάρχει. Είναι μια συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων τομεών δεν θα πρέπει τα GTI και άλλες δομές να θεωρούνται ε, νομικά ε, σαν ε, ακολουθώντα τα καθεστώτα ενός κοινοτικού φορέα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η δυνατότητα δράσης. Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δεχθούν την προσέγγιση αποδοχής του κινδύνου μέσω της ε, ιδιωτικής και δημόσιας ε, εταιρικής σχέσης για να πετύχουν τους στόχους τους. Ξέρουμε ότι είναι εύκολο να το λέει, πιο εύκολο παρά να το κάνει, αλλά η Business Europe βασίζεται στην Επιτροπή σας για να πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, πολύ σαφής, ε, οι ομιλίες σας και μέσα στο χρόνο που σας είχε διατεθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω τον επόμενο ομιλητή, Ρίκ Ντοτριά, εκτελεστικό διευθυντή του Clean Sky, κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν ε, τι είναι ακριβώς αυτό η, ε, το Clean Sky Joint Technological Initiative. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μιλήσω μια άλλη γλώσσα παρόλο που προβλέπετε τα αγγλικά στην επιχείρηση αυτή του Clean Sky, καθαρός ουρανός θα λέγαμε. Προφανώς, το στόχο τη ακρόαση αυτή δεν είναι να σα παρουσιάσω τι λεπτομέρειε ε, τα στοιχεία για το Clean Sky. Άμα θέλετε, μπορώ να επανέλθω κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε να το κάνω αυτό. Παρ' όλα αυτά, εισαγωγικά θα σα ε, υπενθυμίσω κάποια πράγματα για την επιχείρηση αυτή. Το Clean Sky πρόκειται μια τεχνολογική πλατφόρμα που ενώνει το σύνολο των ενδιαφερομένων επιστημόνων, ε, ε, ερευνητών, ε, τεχνολογικών ε, εμπειρογνωμόνων, παραγωγών κλπ. Όσον αφορά το περιβάλλον θέλουμε να μειώσουμε κατά το ίμιση τις, και το θόρυβο και τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι η στόχη του ΑΚΡΕ που προχωράει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το στρατηγικό του τομέα. Το Clean Sky δεν έχει πετύχει ακόμα όλους αυτούς τους στόχους, αλλά επιτρέπει στην βιομηχανία να προχωρήσει αρκετά στις τάξεις του 20-40% χάρη στις ε, δραστηριότητε έρευνα που πραγματοποιούνται. Αναφέρεται στην πραγματοποίηση ε, τεχνολογίας επίδειξης ε, για το θέμα αυτό. Εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα πρωτότυπο δηλαδή. Για να περάσει το πνεύμα του ΑΚΑΡΕ στο λειτουργικό τμήμα, το Clean Sky είναι μια εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ένα Joint Technology Initiative, NGTI. Η κοινή εταιρεία που δημιουργήθηκε με κανονισμό του Συμβουλίου το τέλη του 2007. Βλέπετε εδώ ένα σχήμα του προγράμματος που πραγματοποίησε στο, ε, στις έξι τομείς που καλύπτουν διάφορους τομείς και τύπους αεροσκαφών. Γίνεται επίσης μια τεχνολογική αξιολόγηση, εμείς είμαστε αξιολογητές, βασιζόμενοι στην δυνατότητα να κάνουμε μια πρόβλεψη για την πρόοδο που θα μπορούσε να επιτευχθεί και να εξασφαλίσουμε ότι οι επιλογές που έχουν γίνει είναι σημαντικές. Κάθε ένας από τους ε, άξονες αυτούς βασίζεται σε ένα διτό ηγέτη από δύο leader της ε, βιομηχανίας. Δημόσια χρηματοδότηση τώρα. Έχουμε τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων. Από την μια φορά οι leaders, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, από την άλλη μεριά οι συνδεδεμένοι με τους leaders αυτού, άλλοι βιομηχανίες, ε, έψιλον ε, πανεπιστήμια που είναι τα μέλη αυτά του Clean Sky και είναι δεσμευμένοι για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σήμερα υπάρχουν 84 μέλη συνολικά. Μερικά ενωμένα σε συνδέσμους. Και μια τρίτη κατηγορία που είναι οι εταίροι που επιλέγονται για κάθε προσφορά που γίνεται αυτή τη στιγμή τριμηνία με συμβάσεις ενός έως τριών ετών. Όποιο λέει εταιρική σχέση δημόσιο, ιδιωτικού δημόσιου τομέα σημαίνει κατανομή του ο, κόστους. Και κοινή διαχείριση βέβαια. Υπάρχει ένα governing board, ένα διοικητικό συμβούλιο, όπου εκπροσωπούν 18 βιομηχανικές εταιρείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει δικαίωμα βέτο για τις κύριες αποφάσεις. Η κοινή επιχείρηση έχει ένα εκτελεστικό σώμα επίσης που θα πρέπει να είναι αυτόνομη σε λίγες μέρες. Τώρα εγκαθιδρύεται. Εάν ο Γενικός Διευθυντής, πρέπει ο γενικό Διευθυντής ε, για την έρευνα τη ε, Κομισιόν να επιβεβαιώσει την αξιοθεσία αυτή. Τώρα ήταν η τελευταία διαφάνεια που είχα. Τώρα θα σας τα πω αφήνοντας αυτή τη διαφάνεια μπροστά σας. Τι γίνεται με τα άλλα GTI και όπως είπε και ο Γιάνν Φανεμπίζε πριν από μένα. Πρόκειται για ένα κοινοτικό σώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι υπόκειται στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον κανονισμό που αφορά το προσωπικό. Θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα πλαισίωσης αλλά θα επανέλθω στους δικού που αφορούν το Clean Sky. Είναι γεγονό ότι η δημιουργία του Clean Sky ε, χαρακτηρίστηκε πρόσφατα από έντονη έκφραση ανυπομονησίας από την περιά της ε, βιομηχανίας ε, του κλάδου. Δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπερβάλλουμε στις αντιδράσεις μας, να καταλήξουμε δηλαδή σε συμπεράσματα ει βάρο τη διαχείριση αυτή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Άλλο είναι η φάση της δημιουργίας και άλλη της πραγματοποίησης. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια κοινή πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ θετική για τη συνεργασία αυτή ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και θα πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρει. Είναι προφανές ότι η ορίμαση του Clean Sky επιταχύθηκε πάρα πολύ από πέρσι την Άνοιξη μετά από την πρώτη έκκληση υποβολή προτάσεων με εξέταση των συμβάσεων που σέβονται τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουμένως όσον αφορά τις προθεσμίες. Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων που υπήρχαν σοβαρά για το 2010, επιτάχυνση της πρόσληψης των ατόμων που θα είναι στο ε, στην διοικητική υποστήριξη και γενικότερα η από τις, ε, την Κομισιόν μια ομάδα εργασία που αφορά τα 5 GTI και συμπεριλαμβάνει ε, εκπροσώπους των βιομηχανικών κύκλων και που θα πρέπει πριν από το Δεκέμβριο να υποβάλουν προτάσεις για το μέλλον των εταιρικών αυτών σχέσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον τομέα της έρευνας. Αυτό δείχνει ότι κάνουμε σήμερα και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη για το μέλλον και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάτι θετικό. Θα ήθελα να τονίσω την ε, ποιότητα των σχέσεων μεταξύ της ομάδας του ζήτη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, ορισμένων που προέρχονται από την Κομισιόν κλπ, άλλο που προέρχονται από την βιομηχανία ή από ερευνητικά κέντρα και τους εταίρους τους στην Εκτελεστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη σχέση αυτή και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον κατά τη γνώμη μου. Μια τέτοια κοινή επιχείρηση έχει σαν στόχο στο στρατηγικό ε, τομέα αλλά και στο καθημερινό έργο να συνενωθούν οι, οι εκείνοι που δρούν στον ε, τομέα τον ιδιωτικό και στον τομέα των δημόσιων και στην έρευνα. Αυτό είναι κάτι που αφορά άμεσα τον πολίτη, γιατί πρόκειται για τον έλεγχο των επιδεινώσεων στο κλίμα και της επιδείνωσης όσον αφορά και το θόρυβο. Και αυτό νομίζω δίνει ένα πλήρες νόημα στο Clean Sky. Αυτή η εταιρική σχέση, αν λειτουργήσει, θα ε, πετύχει να προχωρήσουμε πέρα από τους αρχικούς στόχους. Το GTI δεν είναι μία απλή έκφραση της Κομισιόν, διαφοροποιείται από τις διάφορες άλλες ε, υπηρεσίες και όργανα της Κομισιόν. Είναι ένα νέο ζώο, αν θέλετε, που δεν έχει οριστεί ακόμα απόλυτα πράγμα που οφείλεται στις παλιές δυσκολίες, αλλά και που προσφέρει νέες ευκαιρίες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα, ένα περιοριστικό πλαίσιο, αν θέλετε, για το GTI, που μπορεί να να βελτιωθεί με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και τα τελευταία χρόνια. Προσπαθήσανε αυτό το νέο ζώο να προσαρμοστεί περισσότερο στα παλιά που ξέρανε, εις βάρος όμως της λήψη υπόψη του πραγματικού του περιεχομένου. Το θέμα σήμερα δεν είναι γιατί ε, δεν μπόρεσε να προχωρήσει τόσο γλίγορα η εξέλιξη μέχρι στιγμής, αλλά τι μπορεί να την τροχοποιήσει στο μέλλον την εξέλιξη αυτή. Παραδείγματο χάρη θα πρέπει να υπάρξει νέα μέθοδος προσλήψεων που δεν προβλέπεται στον προπολογισμό. η διάρκεια για την υποβολή των, ε, για την απάντηση μάλλον στις κλήσεις για υποβολή προσφορών. Αυτά είναι μάλλον θέματα και στάσεις τόσο πολύ και όχι ε, κανόνων. Ιδίως όμως αυτό που μας ε, δυσκολεύει τη ζωή είναι η διάρκεια για την λήψη αποφάσεων. Γιατί όσο και ανεξάρτητο να είναι το ζητή, εξαρτάται παρόλα αυτά από τη λήψη αποφάσεων σε όργανα της Ένωσης. σαν ε, νεοαφιγμένος ω γενικό Διευθυντή εδώ προερχόμενο από τη βιομηχανία θα, πρέπει να δειχθώ με Δεν έχω ακόμα πολλή εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμω θα ήθελα να σας πω ότι εξεπλάγει πάρα πολύ και θα ακολουθώ να εκπλήττομαι. Η πρώτη πηγή έκπληξη για μένα προέρχεται από το θέμα των ελέγχων για τα πάντα και από την ε, απόρριψη του κινδύνου εκεί είναι νομίζω η βάση η γραφειοκρατία. Κανένα δεν ότι πρέπει να αποφύγουμε τις απάτες ή ότι θα πρέπει να διορθωθούν και να ακυρωθούν τα σφάλματα. Θα πρέπει να εξετάζονται τα θέματα αυτά των ε, δημοσιονομικών ενδεχομένων προβλημάτων, να ελέγχονται οι έλεγχοι. Παρ' όλα αυτό όμως ε, δεν θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος εις βάρος της αποτελεσματικότητας, εις βάρος της ε, λήψη υπόψη του ίδιου του προγράμματος έρευνας. Αυτά δεν ε, οφείλονται μόνο στην Κομισιόν. Καμιά φορά συζητείται το θέμα της ε, καλλιέργειας μιας ατμόσφαιρας μηδενικού κινδύνου. Αυτό οδηγεί βέβαια συν πλήρη αδράνεια. Να υπάρχουν μόνο εγγυήσει και περιορισμός του κινδύνου είναι μια δραστηριότητα που παίρνει όλο το χρόνο και δεν οδηγεί σε δράση. Και είναι πραγματικός κίνδυνος και απειλή για τις μελλοντικές δράσεις. Δίνεται επίσης περισσότερο χρόνο και προσοχή στις διαδικασίες ε, της χορήγησης, ξέρω εγώ, για 10.000 ευρώ ας πούμε, παρά να δούμε ότι οι 10.000 αυτές ε, που δόθηκαν για κάποια δραστηριότητα οδήγησαν σε κάτι θετικό. Αυτός ο μηδενικός κίνδυνος λοιπόν είναι αποτρεπτικός πλήρως. Δηλαδή ο χρόνος που, που σπαταλάτε για να ανοιχτευτεί ε, ένας κίνδυνος για ένα μηδενικό ε, ποσό είναι εις βάρος άλλων δράσεων. Εγώ βέβαια γνωρίζω την αναγκαιότητα του κινδύνου λόγω της προηγούμενης θέσης που είχα. Στη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να διευρύνουμε τον ε, ορίζοντα, χωρίς βέβαια να εγκαταλείψουμε τους ελέγχους, προσπαθώντας όμως να δούμε τι γίνεται με όλους τους τομείς αποτελεσματικότητας. Είναι δύσκολο αυτό. Γίνεται μια προοδευτική προσπάθεια και στην ίδια την βιομηχανία σιγά σιγά. Για τη διαχείριση λοιπόν ενός προγράμματος πολύπλοκου και μακροχρονίου όπως το Sky, η βιομηχανία έχει κάποιες εμπειρίες. Η έννοια του ελέγχου δεν είναι συνεξένη, γιατί βέβαια η βιομηχανία ενδιαφέρει τι γίνεται με τα χρήματά τη. Και το να βρεθούν οι σωστοί κανόνες είναι κάτι που μπορούμε να λάβουμε από κοινό. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι το Clean Sky. Θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική ε, εξέταση λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προθεσμίες και τους συμμετέχοντες. Γιατί δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο business as usual. Ε, ε εφανώνονται μηχανικά ορισμένοι κανόνες που επιβλήθηκαν από την Κομισιόν χωρίς να μπορεί κανένας να αποκλίνει. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας δύσκολος ρόλος, αλλά πάρα πολύ προκλητικός, για να μπορέσει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και κατά δεύτερο το κοινοπληγόρο των κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ξεβρεθούν συγκεκριμένα από κοινού οι διαδικασίες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την ε, ακαμψία των κανόνων, υπάρχει και το πνεύμα με το οποίο εφαρμόζονται αυτοί. Γιατί πολλές φορές ε, μετά από πολλά χρόνια καταλήγουν σε ένα νέο στρώμα ελέγχου, ε, την υπερπιότητα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν. Αυτό το πνεύμα είναι κάτι που δεν βρίσκεται μόνο στην Κομισιόν και στο στους του ίδιου, αλλά είναι και θέμα πολιτικής νομίζω, σε εκείνου που δρούν για την πολιτική δημόσια βούληση. Να μην υπάρχει κανένα σφάλμα, να είναι όλα σύμφωνα με τους κανόνες και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει η διαχείριση μια έρευνα. είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη Θα πρέπει να δεχθούμε ότι τα πρώτα GTI είναι πειραματικού χαρακτήρα, δημιουργούνται οι πρώτες προϋποθέσεις για μεγάλη αποτελεσματικότητα και όπως είπαμε η ίδια η φύση της δραστηριότητας δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. Θα πρέπει με μέτρο να προχωρήσουμε στη μείωση των εμποδίων αυτών. Και για να τελειώνω, το να δεσμευτούμε στην δημιουργία των ε, κοινών ε, σωμάτων αυτών έρευνας, οι κανόνε δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν, αλλά θα πρέπει να είναι πιο καλά και εύκολα εφαρμόσιμοι. Να ανοιχνεύσουμε και να γνωρίσουμε τι κύριε προτεραιότητες. Αυτά είναι νομίζω τα σημεία που ε, δίνουν μια γενική εικόνα για τα πώς θα πρέπει να προχωρήσουν τα GTI και το Clean Sky προτίθεται να κάνει ό,τι θέλει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ακούσαν πάρα πληροφορίες, τα πράγματα έγιναν σαφέστερα, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στους ε, συναδέλφους και Κομισιόν εδώ και το Συμβουλίο, οπωσδήποτε θα μιλήσουν και αυτοί και σας παρακαλώ να αντιδράσετε σύντομα εάν επανέλθετε στι ερωτήσεις σας, γιατί θα έχουμε βέβαια και άλλες ε, ε, ερωτήσεις και θα πρέπει να περάσουμε και στη σύνοψη της κυρίας ΕΚ. Οπότε, πρώτα απ' όλα η κυρία Καρβαλιού έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ε, ομιλητές μας για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Να τονίσω κάτι. Η αξιολόγηση βεβαίως αφορά τις διαδικασίες και όχι το περιεχόμενο της ε, έρευνας και χρειάζεται αυτό το οποίο ακούστηκε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Συμφωνώ πως μια τέτοια κουλτούρα πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να αλλάξει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Αντιλαμβανόμαστε πως ε, πολλές από τις διαδικασίες είναι για προστασία των ιδίων των ε, υπαλλήλων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα είναι πιο σημαντικό και στο μέλλον, δηλαδή να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας Έχουμε πολύ σημαντικό εργαλείο, έχουμε τον 171 και τον 169 ε, για την ε, κοινή εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν που είναι φρικτές διαδικασίες, χρειάζονται 2-3 χρόνια οπότε δεν ε, μπορεί να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας με το 171 και το 169 ως έχουν σήμερα. Πρέπει να απλοποιηθούν αυτά και αυτό αφορά και τον, την αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού. Εν τω μεταξύ συμφωνώ με δύο πράγματα Μπορεί να γίνουν με τον τρέχοντα κανονισμό, δηλαδή να μην πολλαπλασιάζονται τα συστήματα γιατί είναι δύσκολο για όσους κάνουν έτσι να έχουν τόσους διαφορετικούς κανόνες. Δεύτερον, ο χρόνος που θέλει η Κομισιόν για να εξετάσει και να προχωρήσει στις πληρωμές και μετά υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για να απαντήσουν οι εταίροι ε, μέσα σε μέρες ενώ πριν περίμεναν 6 και 9 μήνες για να στείλουν ε, τις ε, εκθέσεις τους. Έχω και άλλα πράγματα, θα τα πω την άλλη φορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορέρα Τεκάμπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους ε, ομιλητές μας ε, για το ότι ήταν θετικές οι παρουσιάσεις τους και ειλικρινείς. Και ήταν βεβαίως και επικριτικές. Δεν ανέμενα τίποτα διαφορετικό. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ αρνητικές για αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να προσθέσω. Το ένα σχετίζεται με τους ε, μικρότερους φορείς καθώς έχουν ακόμα μεγαλύτερο μειονέκτημα όταν είναι αυξημένη η γραφειοκρατία και είναι ακόμη δυσκολότερη για αυτούς η κατάσταση. Και δεύτερον θα ήθελα να επισημάνω εγώ το αρνητικό αποτέλεσμα αυτής της γραφειοκρατίας. Υπάρχει πάνω απ' όλα αβεβαιότητα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απολύτως σίγουροι για το ποιοι είναι οι κανόνες. Στην δε εσωτερική πολιτική μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία μια πολιτική ομάδα ε, ξοδεύει ε, κάποια πράγματα όσον αφορά κάποια ομάδα συμφερόντων και βεβαίως μετά υπάρχουν τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ε, που ερμηνεύουν πολύ στενά την νομοθεσία. Σαν όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν ε, θα μας ε, προξενούσε έκπληξη βεβαίως ε, το ότι καταδικάζεται η γραφειοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποια αυστηρότητα αλλά και σταθερότητα. Αυτό που δεν γίνεται είναι να αλλάζουν συνεχώς οι κανόνες του παιχνιδιού. Οπότε για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Κοιτάξτε, έχουμε ακόμα 4 χρόνια στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 και κάτι πρέπει να γίνει. Και είμαι σίγουρος πως κάτι μπορεί να κάνει το κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να αλλάξει η προσέγγισή μας. Πρέπει να αξιολογούμε την έρευνα με βάση το αποτέλεσμα όχι με βάση τις γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες. Και υπάρχει και η ανάγκη να εκπαιδεύσουμε ε, και τους δικούς μας ανθρώπους να διαχειρίζονται τα επιστημονικά προγράμματα. Δεν φτάνει να έχουμε εξωτερικούς ελεγκτές, πρέπει να έχουμε δικούς μας ελεγκτές που να είναι εξοικειωμένοι με το θέμα. Όπως είπα, είναι δυσκολότερο αυτό για τους ε, για τους μικρότερους φορείς, αλλά το βασικό είναι, όπως είπα, να έχουμε και σωστούς ε, κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους εκείνους που εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους ε, προς ε, τους εισηγητές. Θέλω λοιπόν να σας πω, μας είπαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πράγματα, ε, κυρίως ε, οι παρεμβάσεις ήταν ε, λεπτομερείς και αντιμετώπισαν τα προβλήματα με ένα επικριτικό και κριτικό ίσως πνεύμα που το βρίσκω πολύ σημαντικό. Πρέπει να μιλήσουμε για κάτι όμως το οποίο δεν αναφέρθηκε σήμερα το πρωί. Και κάνω αυτές τις ε, παρατηρήσεις έχοντας κατά νου το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, έχοντας κατά νου το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι εμείς εδώ είμαστε σε, μια, ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αντιμετωπίζει χήμερες με μεγάλη προσοχή κατέγραψα το θέμα της έρευνας σε σχέση με τις ε, βιομηχανικές μονάδες. Έρευνα μεν, αλλά να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό για μας είναι πολύ ενδιαφέρον. Η ευημερία των Ευρωπαίων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της έρευνας. Και εγώ θέλω να κάνω έκκληση σήμερα για το ότι η έρευνα δεν πρέπει να γίνεται χάρη και μόνο της έρευνας. Πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα η έρευνα πρέπει να συνδέεται με χειροπιαστά αποτελέσματα, διότι αλλιώς με κοινέ δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ε, με δραστηριότητες βιομηχανικών μονάδων, οργανικών φορέων. Τελικά η έρευνα που γίνεται προ όφελο ε, της Ευρώπης, αν δεν αποφέρει αποτελέσματα, τότε γιατί γίνεται. Αν ζούσε σήμερα ο Καντ, πού θα ενετάσετε ή το έργο του για την ε, κριτική της ε, λογικής του, μπορούμε να πούμε και για τον Χέγγελ και για τον Σόπενχάουερ. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας αναφέρω, ότι το πανεπιστήμιο, η έρευνα αναμφίβολα πρέπει να ασκούν κριτική, αλλά πολύ συχνά δυστυχώς οι ορισμένε περιπτώσεις δεν είναι χειροπιαστές. Βεβαίως με αυτόν τον τρόπο και η κοινωνία μπορεί να προχωρά σε άλλα επίπεδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την ειλικρίνεια με την οποία οι ομιλητές παρουσίασαν τις παρεμβάσεις τους. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα θέματα. Θα ήθελα να ακολουθήσω τη γραμμή που χάραξα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα δομικά, ε, προβλήματα κοινωνίας, ε, έχουμε μικρές ομάδες, οι οποίες ε, δεν έχουν καθόλου χρόνο στη διάθεσή του, γιατί καλούνται να παρουσιάσουν μία ομιλία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ε, επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν και γραφειοκρατία, δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με την έρευνα. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με πρακτική ε, φύσεως θέματα, θα κάνω κάποιες προτάσεις και θα μου πείτε ποια είναι η δική σας συγγνώμη. Θέλω λοιπόν να σας πω, συμφωνώ με την συνάδελφο από την Πορτογαλία που λέει ότι πρέπει να εκπονήσουμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό για μένα είναι απόλυτα σαφές. Οι προηγούμενοι κανονισμοί Αυτούς τους κανονισμούς τους επιδεινώσαμε εμείς, ε, το Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι αλήθεια ότι έχουμε αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά στη τελική ανάλυση ο καθένας καθέτει τη δική του τροπολογία η μία πιο περιοριστική από την άλλη και τελικά που καταλήγουμε για να πάρει κανείς ένα ευρώ από την Κομισιόν διεξάγονται χιλιάδες έλεγχοι. Πρέπει λοιπόν να συσταθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα μας πει με απόλυτη σαφήνεια από πού μπορούμε να επωφεληθούμε εάν υπάρξει κάποιο είδους ε, φιλελευθερωποίηση. Πρέπει να δούμε τα πράγματα κάτω από αυτό το πρίσμα και θέλω να σας πω ότι και εγώ συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές ότι αν ξεκινάμε ή εφόσον ξεκινάμε από τη δυσπιστία δεν καταλήγουμε πουθενά. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια ε, αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί το ελεγκτικό συνέδριο μας είπε ότι οι ερευνητές ε, πρέπει κάθε πρωί να βρίσκονται στα πανεπιστήμια τους, ε, στα ερευνητικά τους ε, κέντρα, να έχουν παρουσία. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από τους ερευνητές να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό προϊόν Δεν ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ μίλησα με πάρα πολλά στελέχη της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και είπαν ότι όσον αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, η αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει όχι μόνο από ένα, αλλά από πολλά μέρη, από κοινού. Δεν θα πρέπει να ε, δίνουμε την ίδια χρηματοδότηση στους ερευνητές και στους άλλους που διαχειρίζονται θέμα οδοποίησης. Μεταξύ άλλων θέλω να σας πω, έχω κατά νου το ότι πράγματι η Επιτροπή δεν έχει συνηθίσει να λαμβάνει κινδύνους, ε, πόσο μάλλον ε, τα στελέχη από την άλλη, όμως η Κομισιόν δεν συμμετέχει σε εκλογές, ούτε κερδίζει ούτε χάνει εκλογέ. Και α μην ξεχνάμε, η κίνδυνη είναι κάτι το συνηθισμένο στη ζωή μα. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή έχει στελέχη τα οποία δεν γνωρίζουν πώ να διαχειρίζονται καταστάσει. Σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι το Συμβούλιο είναι εκείνο που αποφασίζει για ε, συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, για τεράστια κονδύλια. Και ένα ε, από τα προγράμματα πολιτιστικής εκλονομιάς ε, αφορά την ε, δική μου την πατρίδα. Έχουμε πάρα πολλά ε, έργα που έχουν σχέση με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και πώς είναι δυνατόν τα στελέχη να μην γνωρίζουν ότι αυτά τα θέματα είναι σημαντικά αλλά δεν ε, είναι απαραίτητο για να καταλήξει κανείς σε μια χρηματοδότηση σε ένα και μόνο πρωί να πρέπει να ξανασυζητήσει την, ε, μια συγκεκριμένη όπερα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας δείξω ότι εδώ βλέπουμε υπάρχει ανάγκη δραστηριοποίηση. Ευχαριστώ την Κομισιόν γιατί δείχνει να έχει καλές προθέσεις. Ε, με το Eurostar και το Ευρικά κάναμε καλές εμπειρίες και με τα κοινά ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί προς μια απλουστευμένη ηλεκτρονική καταγραφή. Υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί προς τα εφάπαξα ποσά. Αυτό το δρόμο πρέπει να τον ακολουθήσουμε με συνέπεια. Και όσον αφορά τους ελέγχους, θα πρέπει να μεριμνήσουμε οι έλεγχοι αυτοί να έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση κονδύλιων. Ε, δηλαδή η διοίκηση θα πρέπει σε κάθε έλεγχο που διεξάγει να αναφέρει ποιε είναι οι προτάσει των ελεγκτών έτσι ώστε στο μέλλον να ε, βελτιωθεί το σύστημα. Γιατί υπάρχουν επικαλύψεις ε, στου ελέγχους, παράλληλοι έλεγχοι και όλη αυτή και η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μακρά. Χρειαζόμαστε λοιπόν συντόμευση και αυτό το έδειξαν τα προγράμματα Eurostar και το έβρικα. Ελπίζω λοιπόν στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, όπου ελπίζω να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τα κονδύλια σε σχέση με το 7ο, εκεί λοιπόν στο 8ο να δρομολογήσουμε καταστάσεις, πρωτοβουλίες αν θέλετε, που θα αντιμετωπίσουν κινδύνους και θα είναι και αποτελεσματικές. Η συνάδελφος Ρέρα Μαντουρέλ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ όσους ε, διοργάνωσαν αυτή την ακρόαση. Ε, μία μικρή παρατήρηση μόνο, κύριε Πρόεδρε, παρόλο την εκτίμηση που σας έχω καλό θα ήταν νομίζω εκτός από την κυρία Εκ να υπάρχει και άλλη μια γυναίκα στο Προεδρείο. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ του ε, ομιλητέ για το ότι μίλησαν ξεκάθαρα για ένα πολύ επίκαιρο θέμα για τα πανεπιστήμια και τους ερευνητές μας ε, είναι και εγώ πεπισμένη όπως και οι περισσότεροι νομίζω πως πρέπει να αλλάξει αυτή η κουλτούρα του ελέγχου και να περάσουμε σε ένα σύστημα εμπιστοσύνης. Βεβαίω το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας πω είναι πως ε, το συζητήσαμε αυτό πάρα πολύ κατά την προετοιμασία του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, φαίνεται πως δεν ήμασταν αρκετά επιτυχείς σε αυτό. Θέλω να σας πω πως σημειώσαμε όλα όσα είπατε, ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες, αν και τα γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε αρκετά από αυτά τα ζητήματα. Για να πω πως εγώ τα έχω πει αυτά πολλές φορές απευθυνόμενοι προς την Κομισιόν εντό της Επιτροπής μας. Δύο πράγματα τώρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το πώς ε, λειτουργεί το, το σύστημα που υποτίθεται ότι θα ήταν μια νέα προσέγγιση εντός του προγράμματος πλαισίου όσον αφορά την έρευνα και Δεύτερον, για τις κοινέ τεχνολογικές αυτές πρωτοβουλίες, τα JTI. Εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για ώρες, αλλά να πω πως ε, καλωσορίζω ιδιαίτερα αυτό τα οποία είπε ο κύριος ε, Ντοτρί γιατί στο κοινοβούλιο εμείς πάντα ε, ασχολούμασταν πάρα πολύ με το πρόγραμμα το Clean Sky των καθαρών ουρανών γιατί θεωρούμε πως το JTA μπορεί να μας βοηθήσει να οδηγηθούμε σε SDIT σε συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα αλλά έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την εφαρμογή όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη την διαφάνεια, τους κανόνες συμμετοχής ε, κτλ. Ο κ. Δότρια ανέφερε τα προγράμματα της ε, γραφειοκρατίας, αλλά μας έδωσε μια αισιόδοξη εικόνα του τι συμβαίνει με τις κοινέ αυτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και αλήθεια είναι ότι πολλοί στην Επιτροπή μας έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Δεν το βλέπουμε τόσο καλά όσο ο εισηγητής μας. Π.χ. αν δούμε τον φετινό προϋπολογισμό, πέραν από τα της γραφειοκρατίας, το γενικό επίπεδο εφαρμογή και ειδικά του καθαρού ουρανού είναι πολύ χαμηλό και δεν νομίζω να οφείλεται αυτό μόνο στην γραφειοκρατία. Έχουμε κάποιε αμφιβολίε για το εάν είναι βιώσιμο το σύστημα αυτό για τι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουμε μια διαφορετική συνταγή. Οπότε, για να φύγουμε λίγο από τη γραφειοκρατία, μπορείτε να μας πείτε κάτι επί της ε, ουσίας και όχι μόνο ο κύριος Δοτριά, αλλά και οι υπόλοιποι ομιλητές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για τις ρεαλιστικές ε, προτάσεις ε, του ε, πρόεδρου μας με ικανοποίησαν. Κοιτάξτε, εγώ τους τελευταίους μήνες που ρωτάω σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας γιατί δεν συμμετέχουν, γιατί δεν βρίσκουν πρόσβαση, πάντα μου λένε ότι φταίνε οι κανόνες του προϋπολογισμού. Άλλοι συνάδελφοι νομίζω το ανέφεραν ήδη. Εντάξει, καλός ο έλεγχος, αλλά ο πάρα πολύ έλεγχος δεν είναι καλύτερος. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος γιατί έχουμε μια ευθύνη για τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά νομίζω πως πρέπει να οδηγηθούμε έτσι και σε μια λογική σε ένα μέτρο για να μην εμποδίζουν πάρα πολύ την πρόσβαση οι κανόνες. Έχω τώρα εγώ τρεις ερωτήσεις ε, για τους ε, εκπροσώπους εδώ πέρα. Δύο απευθύνονται στον κύριο Φαντεμβίζεν, τον εκπρόσωπο του Business Europe. Ο κύριος Πάλεσεν ε, είπε πως κάποιους από τους κανόνες που έχουν γραφτεί ακριβώς για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη ως εκπροσώπου της Business Europe. Και κύριε Βίζεν, να ρωτήσω και σας, εάν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ποσοστό συμμετοχή σε αυτά τα ερευνητικά μέσα, αν έχουν επιτευχθεί. Και το τρίτο ερώτημα απευθύνεται σε όλους σας. Ε, ο κύριος Χάλ έκανε την πρόταση μια στρογγυλής ε, τραπέζης ε, μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και ειδικά στην Επιτροπή μας για να επεξεργαστούμε τους μελλοντικού κανόνες. Συμφωνείτε και οι υπόλοιποι με αυτή την ιδέα. Ευχαριστώ η κυρία Τόια. Grazie Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι, τους ομιλητές για τη σαφήνεια με την οποία μίλησαν και για τις προτάσεις που κατέθεσαν και τις αναλύσεις που μας παρουσίασαν. Νομίζω ότι πέρα από κάθε αμφιβολία κατέστη σαφές ότι σήμερα υπάρχει δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτό που είναι το περιεχόμενο ενός προγράμματος και την αξιολόγηση του αποτέλεσματός του. Αυτά αφενός και αφετέρου τη συγκέντρωση των κονδυλίων, του χρόνου, της γραφειοκρατίας αλλά και των προτεραιοτήτων για την διαδικασία, για τους κανονισμούς, για τα διοικητικά έγγραφα, για την αξιολόγηση του κόστους κτλ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ανατροπή αυτό που λέμε μεσ, μέτρου, μάλλον μέσου και στόχο. Ο στόχος γίνεται μέσο και αντίστροφα. Κατόπιν τούτου, αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί και ε, όλοι τα έχουμε ακούσει στις ε, χώρες μας, όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στο να αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία για να ε, καταλήξουμε σε μία συγκεκριμένη ανάλυση. Ποιος θα αναλάβει εγώ λοιπόν απευθύνομαι σε εσά. Αν πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την αναλογία μέσου και στόχου για πολλά θέματα, όπως είναι κάνει συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αν το κάνουμε αυτό, εσείς τι προτείνετε τελικά, εφόσον μειωθεί το διοικητικό άγχο και η έλεγχη, θεωρείτε ότι πραγματικά θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και πώς πρέπει να εξοπλιστούμε για να επιτύχουμε το στόχο μας. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα σε μια εθνική πρωτοβουλία στη δική μου τη χώρα, δηλαδή εκεί εκπροσώπησα το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν μια συνεδρία αφιερωμένη στην έρευνα. Παρίστατο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, δηλαδή η ανώτατη αρχή. Και αυτή η μερίδα οργανώθηκε από ε, τους, τον, την Ένωση των Βιομηχάνων. Και εκεί βεβαίως αναφέρθηκε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Ευρώπη στην έρευνα. Κάτι που θέλω να πω, απευθυνόμενοι στον πρώτο ομιλητή. Κοιτάξτε, το να συγκεντρώνονται όλοι οι διαγωνισμοί, να υπάρχει συγκεντρωμένη προκήρυξη διαγωνισμών, εγώ κατά την άποψή μου θεωρώ ότι δεν είναι καλό. Θεωρώ ότι η προκήρυξη διαγωνισμών ε, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επικρατεί και απόλυτη σαφήνεια. Δηλαδή οι ερευνητέ να γνωρίζουν πότε θα προκηρυχθεί ο τάδε διαγωνισμό και πότε ο δίνα. Το να ξέρει κανείς ότι όλα θα παρουσιαστούν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό κατά την άποψή μου δημιουργεί σύγχυση και γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουμε μεγαλύτερη σαφήνεια περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ο κύριος Τσουκαλάς παρακαλώ. Okay. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους και ομιλητές για τις πολύ σαφείς θέσεις τους. Ε, είναι απογοητευτικό ότι μολονότι τα σημάδια του τι θα συνέβαινε στο 7ο πλαίσιο ήταν από το 2005 γνωστά. Να σας θυμίσω την, ε, το ενδιάμεσο report COC που προανήγγειλνε ήδη τις ε, δυσκολίες της γραφειοκρατίας Το περιβάλλον που μας περιέγραψαν οι ομιλητές σήμερα δείχνει ότι υπάρχει, όπως ανέφερε ο κύριος Χαλ, υφέρποντα συστημικά προβλήματα. Ε, το Πολυτεχνείο μας είπε ο κύριος Παλένων ότι δεν δίνουμε προσοχή στο ερευνητικό αποτέλεσμα και ενδιαφερόμαστε, επικεντρωνόμαστε στη γραφειοκρατία. Και τέλος ακούστηκε αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, ότι υπάρχει δυνατότητα υποκειμενικής ερμηνείας ε, των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των διαφόρων κανόνων που επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία από αρμοδίους ή αναρμοδίους της ε, Κομισιόν. Κοιτάξτε, η των διαφορων κανονων που επιδεχονται διαφορετικη ερμηνεια απο αρμοδιους η αναρμοδιους της κομισιον κοιταξτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η στρατηγική της Λισαβόνας στους σταθέντες στόχους φαίνεται λίγους μήνες πριν από το 2010 να έχει αποτύχει. Μία συνιστόσα της αποτυχίας ή της έλλειψης της επιτυχίας που θα θέλουμε σε αυτή τη στρατηγική φαίνεται να είναι η γραφειοκρατία. Όχι ότι δεν υπάρχει και σε άλλες χώρες γραφειοκρατία. Είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγο καιρό να ακούσουμε τον κύριο Άλαν Λέσνερ τον εκδότη του Science στην εναρκτήρια διάλεξη του GRC να παραπονείται ότι το 42% του ελεύθερου χρόνου των Αμερικάνων ερευνητών πηγαίνει σε γραφειοκρατικές και διηγητικές ενασχολήσεις και ότι μία μόνο από τις πέντε αιτήσει που κάνει για εξωτερική χρηματοδότηση πετυχαίνουν. Εκείνο που με απασχολεί κύριε Πρόεδρε, όπως είχα και την ευκαιρία να σας πω και σε άλλες φορές, είναι ότι όλες οι παγκόσμιες έρευνες που δημοσιεύονται, είτε αυτές είναι η πρόσφατη μελέτη που παραγγείλαμε το 2008 για τις τάσεις το 2025, όσο και η αντίστοιχη μελέτη των Αμερικανών για τις παγκόσμιες τάσεις του 2025, δείχνουν ότι η Ευρώπη χάνει το παιχνίδι του ανταγωνισμού στο στάδιο του R&D. Έχουμε καλές επιτυχίες κάπου, έχουμε συνολική αποτυχία γενικώ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να μας απασχολήσει και πέρα από το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της γραφειοκρατίας που ώρες ώρες μου θύμιζε δίκη του Κάφκα ή μου θύμιζε άρωμα γραφειοκρατίας των ημερών του Μπρέσνιεφ έτσι όπως περιγραφόταν από τους κυρίους ομιλητές ε, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που είπε μία συνάδελφος το κλίμα της καθολικής δυσπιστίας που απορρέει από τους κανονισμούς μας πρέπει να υποκατασταθεί με ένα κλίμα διαφάνειας όπου οι δύο συμβαλόμενοι θα έχουν εμπιστοσύνη ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα Παρόλο που έχουμε διαπίεση χρόνου, να δώσω το λόγο στον κύριο Κίρτζελμπον, τον εκπρόσωπο τη Σουηδική Προεδρία. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ που είναι σήμερα μεταξύ μα. Ίσως θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους για την τόσο επίκαιρη και ενημερωτική μήνυ ακρόαση. δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει, το μίνι ακρόαση δεν καταλαβαίνω γιατί. Μεγάλη ακρόαση μου φαίνεται εμένα. Βέβαια, αυτά όλα δεν θα ολοκληρωθούν ε, κατά τη διάρκεια της ε, Σουηδικής ε, Προεδρίας. Ε, δεν μπορώ παρά να σας κάνω άρα κάποιες προβλέψει για το αποτέλεσμα σε σχέση με την απλούστευση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω και κάποιε σκέψει όσον αφορά τις επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών αποτελεσματών σε σχέση και με την ε, συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πρώτη πρόβλεψη. Θα υπάρχει έντονη υποστήριξη, κατά τη γνώμη μου, των σχεδίων που έχει προαναγγείλει η Κομισιόν του χρόνου να κάνει μια ανακοίνωση για απλούστευση. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ταυτόχρονα, δεύτερη πρόβλεψη είναι αυτή, θα μπορούσα να πω ότι οι προσπάθειες που ε, σκιαγραφεί η Κομισιόν και το Συμβούλιο, και θα επανέλθω σε αυτές αργότερα, απαιτούν για την εφαρμογή τους πάρα πολύ έντονη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Γιατί εδώ αναφερόμαστε στις ιδιαιτερότητες της έρευνας. Ας μην έχουμε αυτά πάντως πολλοί συνάδελφοι σε πολλούς πολιτικούς ε, ε τομείς ε, θα αρχίσουν να αντριχιάζουν ακούγοντας αυτά που λέμε. Και ιδίω ε, επειδή από ένα τομέα κάτι τέτοιο είναι μεταδοτικό σε άλλου τομέα, θα υπάρχουν λοιπόν αντιδράσει και αντιεπιθέσεις όταν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από την άκουσα αυτή η προσέγγιση που βασίζεται σε εμπιστοσύνη και αποτροπή της δυσπιστίας. Ελπίζουμε ότι δεν θα οδηγήσει σε αυτό που γνωρίζουμε ότι όδινε ε, ε και σκέτη και μη. Ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει πραγματικά, πρακτικά αποτελέσματα. Και γιατί. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ο καθορισμός των κανόνων, αλλά και η εφαρμογή και η διαχείριση αυτών των κανόνων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό σχετίζεται με διαχείριση σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων και των επιπέδων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα μηνύματα που αποστέλουμε προς την Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι το εκτελεστικό όργανο υπεύθυνο για την εργασία αυτή. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το σύνολο των κανόνων και η μορφή των κανόνων είναι σημαντική για εκείνους που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτό, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι μόνο θέμα ερευνητικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε αυτούς, να πείσουμε και τους συναδέλφους σε άλλους τομείς πολιτικής, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, όσον αφορά την ανάγκη να κοιμηθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ελπίζω ότι έγκαιρα του χρόνου θα δούμε μία ανάλυση κόστος ωφελίας όσον αφορά τους ισχύοντες σήμερα κανόνες για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλώς θέλουμε να εξετάσουμε κάθε λεπτομέρεια αλλά βασίζεται και στη φιλοδοξία να υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο τόσο πολύπλοκο αυτό θέμα. Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε και εδώ παρουσιάζω κάποιες σκέψεις ε, πάνω σε αυτά που σας είπα. Θα πρέπει, λέω, να βασιστούμε ίσως στην ιδέα του Christopher Hall να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και αναφέραμε εδώ στα τρία κύρια σώματα υπεύθυνα, που είναι υπεύθυνα, αυτό ίσως θα οδηγήσει ίσως σε έναν κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς στη συζήτηση και την εφαρμογή των πολιτικών για την απλούστευση. Γιατί αυτό δεν είναι ένα σχέδιο για έξι μήνες, αλλά μάλλον για έξι χρόνια. Και θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση για όλο αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ρωτώ τώρα την ε, Κομισιόν. Κυρία Τελατόρε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι σύντομη γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πια χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε και εμείς σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ακρόαση, ε, πολύ χρήσιμη για τη δουλειά της Κομισιόν. Η απλούστευση για μας είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι θέμα επιβίωση και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν δεσμεύεται γι' αυτό το θέμα είναι η πρόθεση της ε, Κομισιόν την επόμενη άνοιξη να καταθέσει μια ανακοίνωση σχετικά με την απλούστευση. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, το κολέγιο των, το Σώμα των Επιτρόπων σύντομα θα πρέπει να ανανεωθεί και ε, το θέμα του προπολογισμού είναι ένας βασικός στόχος σε αυτή τη φάση, όπως και η απλούστευση. Και αυτός ένας άλλος βασικός στόχος. Ε, όπως αναφέρθηκε και εδώ, είναι θέμα ισορροπίας, ε, θέμα δόσεων, ε, που, πόσο θα, ποια δόση, ποιο, ποιο κομμάτι θα αντιστοιχεί στην απλούστευση, ποιο άλλο κομμάτι στην χρηματοδότηση. Ας μην ξεχνάμε ότι στη δουλειά μας υπάρχει πάντα και ένα ποσοστό 5% λάθους. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που έχουν ε, εντοπιστεί. Παραδείγματος χάρη το θέμα των εφάπαξ ποσών. Ε, το ελληνικό συνέδριο παρεμπιπτόντος ε, τάσσεται αναπιφλέκτα υπέρ των εφάπαξ ποσών οι ελλείψεις ε, στην εφαρμογή της απόφασης Κομισιόν για τη χρήση του μέσου κόστους ε, προσωπικού και αυτό πάλι είναι θέμα ισορροπίας. Και βεβαίως ε, η ισορροπία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο όπου θα πρέπει να αλλάξει εφόσον αλλάζουν και οι παράμετροι. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου καλεί την Κομισιόν να μην υπολογίζει το κόστος ε, με βάση το πρόγραμμα υπαριθμών 6. Εμείς προσπαθούμε να δούμε ε, πώς αυτό το ψήφισμα θα το εφαρμόσουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι το Κοινοβούλιο ε, χαιρέτησε τη μείωση του ποσοστού ε, λάθους ε, στις, στα προγράμματα που ελέγχονται από την Κομισιόν κατά 8 περίπου της το 2006, άρα δηλαδή φτάνουμε στο περίπου 2% το 2007. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό έγινε μέσα από την εφαρμογή, των, την εκτέλεση των εκστρατιών ελέγχων. Η Κομισιόν ε, δέχτηκε πάρα πολλές κατηγορίες σε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα με απόλυτη σαφήνεια να σας πω ότι η Κομισιόν επουδενή δεν έχει τροποποιήσει την ερμηνεία των κανονισμών. Το θέμα είναι ότι η Κομισιόν έχει ενισχύσει αυτούς τους ελέγχους και Όσο περισσότερο δει κανεί ε, τα προγράμματα, θα δει ότι τόσο πιο, πολύ, τόσο πιο πολλά θέματα τίθενται επιτάπητο. Θέλω επίση να πω ότι ακόμα και αν η Κομισιόν κατέβαλε ποσά και υπογράφηκαν αυτέ οι καταβολέ από δύο υπαλλήλου, όπω πολύ σωστά αναφέρθηκε, η συμφωνία προβλέπει ότι υπάρχει μία περίοδος ανάκλησης, γιατί πολλοί από τους ε, από θέματα που εντοπίζονται ως λάθη μπορούν να εντοπιστούν μόνο με επιτόπιους ελάχου. Άρα δηλαδή η Κομισιόν ε, δεν ε, ανακαλεί, απλά η Κομισιόν σε ορισμένες περιπτώσεις έχει βρει και επιπρόσθετα παραστατικά. Αυτό ήθελα απλά να προσθέσω. Και για να ολοκληρώσω, επιβεβαιώνω την δέσμευση της Κομισιόν να προχωρήσει στο θέμα της απλούστευσης, γιατί σας λέω, για μας είναι θέμα επιβίωσης και όπως είπαν και ορισμένοι ομιλητές, είναι θέμα αξιοπιστίας και θέμα υγείας της ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας. Υπολογίζουμε στη δική σας την υποστήριξη για μελλοντικές προτάσεις της Κομισιόν, τόσο όσον αφορά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, όσο και ε, τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Και βεβαίως ε, εμείς επιθυμούμε ε, να μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε άλλο κανόνα που θέλετε εσείς να θέσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο να πω είναι κάτι επί της αρχής περισσότερο, αλλά θα ήθελα να πω κάτι ξεκάθαρο. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όχι μόνο να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο θέλει η Κομισιόν, αλλά εάν θεωρούν πως κάτι χρειάζεται βελτίωση θα αναζητήσουμε και εναλλακτικέ. Αυτή είναι και η αποστολή μας τώρα. Θα ήθελα να ξαναδώσω τον λόγο ξανά στους ομιλητές μας. Η... κύριος Φων σας παρακαλώ μια μικρή παράκληση, αν μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα αυτές τις πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Στηρίζω πολλές από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των βουλευτών. Η κυρία Ρέιρα Μαδουρέλ ανέφερε πως ε, και στην συζήτηση του προγράμματος 7 τα είχαμε συζητήσει αυτά και αναζητήσαμε βελτιώσεις, πράγματι. Ήδη το 2005 και το 2007 εδώ στο Κοινοβούλιο είχα αναφέρει την έλλειψη εμπιστοσύνης και ανοχής για τον κίνδυνο, αλλά νομίζω πως δεν είχαν ορισμάσει οι συνθήκες. Αλλά ακούγοντας τα σημερινά σχόλια νομίζω μπορούν να γίνουν αλλαγές. Η ήταν μετά κάποια ερωτήματα που απευθύνονταν σε μένα συγκεκριμένα από τον κύριο Μπουτικόφερ και αφορούσαν τις ε, διατάξεις για τις δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι από τα πανεπιστήμια ότι δεν είναι τόσο ελκυστική για τους ερευνητικούς οργανισμούς για να δράσουν. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέει ο συνάδελφος, από την άλλη μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληρώσει και αναμένουν κάποια αποτελέσματα. Τώρα δεν ξέρω απ' έξω την διατύπωση του άρθρου 51, 52, 53 για τους κανόνες συμμετοχής, η Κομισιόν μάλλον θα ξέρει, ελπίζω, αλλά νομίζω πως υπάρχει αρκετό εύρος ε, για τα δικαιώματα πρόσβασης έτσι ώστε να συνεχίζει την έρευνα ο ερευνητικό οργανισμό και να δώσει βεβαίω και στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αυτό για το οποίο πλήρωσαν. Το άλλο ερώτημα, οι στόχοι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή 15% στο πρόγραμμα πλαίσιο, εάν είναι ρεαλιστική, είναι σε κάποια μέρη, αλλού όχι, γιατί δεν υπάρχουν τόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που θα είχε νόημα η συμμετοχή τους και βέβαια πρέπει να μιλάμε πάντα για συμμετοχή με νόημα για όλους τους συμμετέχοντες. Και το τελευταίο ερώτημα που απευθύνονταν σε όλους μας από τον κύριο Μπουτικόφερ ήταν το εάν υποστηρίζουμε την ιδέα του Κρίς Χάλ για μια στρογγυλή τράπεζα για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα του μέσου κόστου. Ναι, βεβαίως την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι πολύ καλή ιδέα αυτή η στρογγυλή τράπεζα, την υποστηρίζουμε. Κοιτάξτε, έτσι όπως πήγε η συζήτηση φαίνεται πως μπήκαμε στις διαδικασίες στη γραφειοκρατία ε, εκεί που και πράγματι χρειάζεται μια συντόμευση, μια απλοποίηση. Δεν έχω αντίρρηση. Τώρα δεν θέλω να περάσουμε στις λύσεις εάν το λένε αυτό οι πολιτικοί μας φαντάζομαι πως αναμένουν από τους υφισταμένους τους να το κάνουν. Όταν κάποιος ε, ασκεί ηγεσία δεν είναι ανάγκη να τα κάνει όλα μόνος του. Υπάρχουν άνθρωποι για να τα κάνουν αυτά. Όταν κάποιοι στο κορυφαίο επίπεδο θέλουν να λυθεί κάτι, νομίζω αυτό πρέπει να αρκεί. Κατόπιν. Το ζήτημα ελέγχου έναντι της εμπιστοσύνης. Φοβάμαι από αυτά τα οποία άκουσα σήμερα, ίσως θα κάνουμε το επόμενο λάθος και θα έρθουμε σε 10 χρόνια και να πούμε πως δώσαμε πολύ εμπιστοσύνη και τώρα κάνω ο καθένας ό,τι θέλει και δεν είχαμε και αποτέλεσμα. Είναι όπως όταν μπήκα εγώ στο ντους σήμερα το πρωί, δεν θέλω ούτε να καώ από το νερό, που είμαστε τώρα δηλαδή, εάν θέλετε, στη φάση του ελέγχου, αλλά ούτε και να βγει παγωμένο το νερό. Ένα χλιαρό. Μία μέση οδός δηλαδή μεταξύ ελέγχου και εμπιστοσύνης, γιατί και πλήρης ε, εμπιστοσύνη, αντιλαμβάνεται τι, σε τι κατάχρηση θα οδηγήσει. Οπότε δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε κανένα άκρο. Αλλά τώρα είμαστε στο άκρο του ελέγχου. Η άλλη ε, διάσταση. Ελέγχουμε το λάθος πράγμα. Ελέγχουμε τα χρήματα. Που, εντάξει, καλό είναι. Αλλά δεν ε, ελέγχουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Τι είναι σημαντικό λοιπόν. Όταν οι ελεγκτές κανονίζουν τους ελέγχους τους, κρίνουν την πιθανότητα του να πάει κάτι λάθος, την ε, σημαντικότητα και το μέγεθος. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εδώ πέρα. Πιθανότητα, σημαντικότητα και μέγεθος. Και το ίδιο πρέπει να γίνει και από το ε, πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να μαγνηθούμε από τον υπερβολικό έλεγχο προ την κατεύθυνση, χωρί να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Προ την εμπιστοσύνη, χωρί να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Οπότε, πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την χρηματοδότηση ή για το αποτέλεσμα. Πάλι πρέπει να βρούμε το σημείο ισορροπία μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα τη κυρία Ζεγιά Μάντζουλα για το Clean Sky. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Clean Sky είναι ένα πρόγραμμα έρευνας που έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί συντονίζονται από τους μεγάλους ε, βιομηχανικούς ε, παίκτες στον τομέα της ενεργειακής για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί μετά να μεταφερθεί σε εμπορικά προϊόντα. Δεν σε τίποτα να υπάρχουν θαυμάσιες ε, τεχνολογίες που μειώνουν το θόρυβο ή τις εκπομπές διοκτήτου του άνθρακα, εάν δεν είναι εφαρμόσιμα και ανταγωνιστικά στον εμπορικό τομέα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η δομή του Clean Sky που απαιτεί η ατζέντα που προβλέπει η Κομισιόν να αφιερώνει χρόνο όχι μόνο στην γραφειοκρατία αλλά και στον έλεγχο του περιεχομένου. Όσον αφορά το πώς ε, γίνεται καθημερινή εργασία. Δεν αναφέρθηκα. Άρχισε όμως από τα μέλη του Clean Sky ήδη τα μέσα του 2008. Προφανώς δεν υπάρχουν ακόμα θεαματικά αποτελέσματα. Αλλά οι εργασίες γίνονται φυσιολογικά θα έλεγα παρόλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν για λόγω της δυσκολίας της εφαρμογής. Θα ήθελα να τονίσω ότι τον Ιούνιο έγινε η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για 70 περίπου θέματα. Η διαδικασία επιλογής έγινε το Σεπτέμβριο με απόλυτα διαφανή τρόπο. Υπάρχει νομίζω κοινή βούληση όλων των εμπλεκομένων μελών να διατηρηθεί μια διαδικασία αδιαφάνειας και πρέπει να το πούμε ότι θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά αυτοί οι μέθοδοι που και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικέ. Τώρα τελειοποιούνται συμβάσεις για περίπου 100 νέους εταίρους και από εκεί και πέρα, τρίμηνο, θα υπάρχουν νέοι εταίροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια κλπ που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Και θα ήθελα την ευκαιρία να αναφέρω ότι τα στατιστικά τη πρώτη αυτή υποβολή προτάσεων καταδεικνύουν ότι το σύνολο των επιλεγμένων εταίρων το 1 τρίτο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράγμα που μου φαίνεται πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω και εγώ τρία σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σας πω, ε, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό που και εσείς στηρίξατε, να υπάρξει μια στρογγυλή τράπεζα ανάμεσα σε, στους τρεις, ε, τρία, στα τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρξει ένα συμφωνία επί του μελλοντικού προγράμματος πλαίσιο. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει. Δεύτερον, Το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από το ότι η προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου για τους ελέγχους είναι υπερβολική, κατά τη γνώμη μου. Αξίζει να έχουμε κατά νου ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογίας και κάθε κράτος έχει το δικό του το ελεγκτικό συνέδριο ή αυτό που αντιστοιχεί με ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ τις τελευταίες εβδομάδες προσπάθησα να ενημερωθώ λιγάκι και δεν άκουσα κανένα κράτος όπου το ελεγκτικό συνέδριο να είναι τόσο επικριτικό και αυστηρό για τη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων έρευνας και εγχολογίας όσο είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ίσως εσείς ως ευρωβουλευτές μπορείτε να το κοιτάξετε λίγο στις πατρίδες σας για να δείτε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει πουθενά ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο στην Ευρώπη. Τέλος, δεν πίστευα ότι θα ακούσω την κυρία Ντελατόρα να ε, λέει ότι η Κομισιόν ε, πρόκειται να θεωρήσει το κόστος. Εγώ όμως θέλω να της πω το Αν κάτι μοιάζει, τρέχει, ε, έχει την εικόνα του σκύλου, ε, λυπάμαι πάρα πολύ, είναι τελικά σκύλος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εκ θα πάρει το λόγο που άκουσε για πάρα πολύ, υπομονετικά. Πρώτα απ' όλα να σα πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ακρόαση που οργανώσετε. Άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Εκ. Κοιτάξτε. Εγώ ήμουν άτομο που έχει γράψει τέτοιε αιτήσει, έχει υποβάλει αιτήσει, έχει λάβει χρηματοδότηση, έχω υποστεί ελέγχου αρκετού. οπότε ξέρω ακριβώς τι σημαίνει συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα. Τώρα, για να επανέλθουμε στη γενική εικόνα, μιλάμε για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Μιλάμε για το πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί με άλλες περιοχές του κόσμου και πώς θα δημιουργηθούν δουλειές και πλούτο στην Ευρώπη. Και όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό μέλλον πάντα αναφέρουμε την έρευνα και την καινοτομία ως ε, βασικό μέσο. Γι' αυτό πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική γιατί μιλάμε και για χρήματα των φορολογουμένων όπως αναφέρθηκε. Ε, τώρα γνωρίζουμε πως το σύστημα δεν είναι όσο, τόσο αποτελεσματικό όσο θα μπορούσε. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό. Σε 10 χρόνια θα έχουμε πάνω από 600.000 600 Κινέζους έρευνητές ε, που θα έχουν αποφοιτήσει στο εξωτερικό και γύρω στους 300.000 στην Ινδία. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και βεβαίως αυτό το οποίο έχουμε εμείς στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και στις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες είναι ε, αν θέλετε, κάτι ανάλογο με την προσελήνωση και δεν θέλουμε να κολλήσουν οι αστροναύτες στα γραφειοκρατικά. Νομίζω ε, επισημάνθηκαν αρκετά προβλήματα και η φήμη μας βεβαίως δεν είναι μόνο ανταγωνιστικότητα. Όπως είπε και ο κύριος Πάλεσεν, μέχρι στιγμής είχα, έχουμε 160.000 ανθρώπους που έχουν ζητήσει χρηματοδότηση. Εάν η φήμη μας είναι πως είναι δύσκολα τα πράγματα ή αδύνατα, διακινδυνεύει το καλό όνομα το δικό μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Εάν δούμε λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν, ακούσαμε από την ΕΑΡΤΟ, την Ένωση αυτή, πως πολλοί από τους ε, μεγάλους χρηματοδότες έχουν ε, προβλήματα, τα ερευνητικά Ινστιτούτα δηλαδή, και είναι φρικτό να ακούμε πως ε, τώρα έχουν πάει τα ερευνητικά δικαστήρια την Κομισιόν στο δικαστήριο για τον έλεγχο. Ε, περιπτώσεις 6-10 ε, ετών είναι έσχος να ακούμε πως μπορεί κάποιος να δεχτεί μέχρι και 6 μάλλον να δεχτεί ελέγχους 6 και 8 χρόνια μετά το τέλος του έργου. Μιλάμε για ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο. Δεν είναι πίνες. Δεν καταδικάζεται κανείς διαβίου. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πάλισαν. Πράγματι πρέπει να ληφθούν κάποιες στρατηγικές αποφάσεις που θα συνεισφέρουν στο να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Συμφωνώ με την προσέγγιση του 50%. Και η δική μου εμπειρία από τη βιομηχανία και το πανεπιστήμιο αυτή είναι. Και εάν δείτε την προθεσμία των 60 ημερών, νομίζω θα τη δείτε στο μέλλον από την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Η άποψη τώρα της ε, βιομηχανίας. Η επιθυμία όλων των πολιτικών ομάδων εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη συνεισφορά και συμμετοχή από τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το να βλέπουμε ότι αποσύρεται από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα η βιομηχανία είναι καμπανάκι που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Τώρα για τις ε, κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Εγώ το παίρνω πολύ σοβαρά και βλέπω πως το ίδιο κάνει και η βιομηχανία και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί αν δείτε το, τον καθαρό ουρανό και τους στόχους του σε λίγα μόνο χρόνια, λύνει το, τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε στην ευρωπαϊκή αεροπορία. Και αν θέλουμε να έχουμε αεροναυτικό κλάδο, Πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα σε 3-4 χρόνια. Και είμαστε τώρα μόλις ένα μήνα πριν την Κοπενχάγη που επίσης ε, πρέπει να μας απασχολήσει αυτή τη βιομηχανία. Οι κοινέ αυτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες υποτίθεται ότι θα ήταν απλές και ανοιχτές και διάφανες. Και όταν βλέπω ότι πάνε σε άλλη κατεύθυνση... Ε, ανησυχώ, εν πάση για να μην πω τίποτα άλλο. Και νομίζω πως θα επανέλθει η Επιτροπή. Τώρα, πώς θα έρθει η αλλαγή. Έχουμε τρία θεσμικά όργανα. Το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ξεκίνησε. Είναι σε καλό δρόμο με αυτή την ακρόαση. Θα συζητηθεί αυτό στο μέλλον. Θα συζητήσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Έχουμε οπωσδήποτε τα ζητήματα προπολογισμού θα δούμε τις συζητήσεις για τη στρατηγική της Λισαβόνας ή τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα σε λίγες εβδομάδες και προβλέπω εγώ ότι θα υπάρξουν ρήτρε από την Επιτροπή μας στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην ευρωπαϊκή έρευνα. και θα είναι μέρος των συμπερασμάτων για τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό η Κομισιόν. Ξέρω πως ε, και ο Επίτροπος ε, είναι στον ίδιο δρόμο με μας. Ε, αναμένουμε την ανακοίνωση για την απλοποίηση. Είδαμε σήμερα πως πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν και μπορεί να γίνουν ήδη εντός του εβδόμου προγράμματος πλαισίου. Προβλέπουμε μια καλή ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα αυτό και θα συνεχίσουμε την ε, συνεργασία. Είχαμε κάποιες προτάσεις και κάποια επιτεύγματα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν για την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι πολύ σημαντική. Τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο, ελπίζω τα συμπεράσματα να περιέχουν κάποιες σχετικές διατυπώσεις. Ακούσαμε πως υπάρχουν ελπίδες, γνωρίζω πως ε, ο εκπρόσωπος εδώ του Συμβουλίου είναι από τους συντάκτες του κειμένου. Αναμένω λοιπόν κάποια σοβαρά λόγια σχετικά και θέλω να σας ζητήσω να το θέσετε αυτό το θέμα και στους Υπουργούς Οικονομικών γιατί έχουν ευθύνη όπως είπαν πολλοί ομιλητές, θα το θέσουμε εμείς και σε άλλες επιτροπές. Και τέλος, για να τελειώσουμε την ακρόαση, ευχαριστώ τους ομιλητές μας, ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές, ε, τους ακροατές, την γραμματεία. Εγώ όταν το είχα προγραμματίσει ο τίτλος ήταν «Θα σκοτώσει η γραφειοκρατία την ευρωπαϊκή έρευνα» και είχα ένα ερωτηματικό. Νομίζω τέλος πάντων ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Two minutes, well, one minute, and then we point another point. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Thank you very much. Thank you very much. Absolutely. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα παρακαλώ λίγο γρήγορα. Για να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο.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 Συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. the most important person we're searching for now. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ημερησία μας διάταξη. Πρόκειται για το θέμα του διαλόγου μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Μια νέα εταιρική σχέση για τον εξορισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ σύντομη εισαγωγή σήμερα. Η εισηγήτρια η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ θα μας κάνει μια παρουσίαση και εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω εάν αρκεστούμε σε αυτήν την εισαγωγή για να προφτάσουμε να εξετάσουμε και το άλλο θέμα γιατί έχουμε καλέσει πάλι. Κυρία Μαντουρέλ, δική σας ε, σειρά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Πρόκειται για τον διάλογο πανεπιστημίων επιχειρήσεων, ε, μια καινούργια σχέση που προκύπτει και για να δοθεί, ε, δοθούν, δοθούν σάρκα και οστά στην παλαιότερη πρόταση Κομισιόν ε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια σχέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις και αυτό έχει ως στόχο να ικανοποιούνται ταχύτερα οι επιθυμίες της αγοράς αλλά και ε, να μπορεί κανείς να αποκτήσει με μεγαλύτερη ευκολία επιστημονική γνώση. Τον Φεβρουάριο του 2008 υπήρξε μία πρώτη συνεδρίαση υπό το πρίσμα της ε, ε, οικονομικής ύφεσης. Ε, αργότερα ακολούθησε μία δεύτερη συνεδρίαση και από όλα αυτά φάνηκε πόσο σημαντικό είναι το πνεύμα της ανακοίνωσης, δηλαδή το ότι πρέπει κανείς να δράσει με ταχύτητα. Εμείς τώρα λοιπόν αναλύουμε αυτή τη δουλειά, τη δουλειά του φόρουμ και πρόκειται κυρίως ε, για τις ε, προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρόκειται επίσης και για τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις που και αυτή χρήζει βελτίωσης. Ε, υπάρχουν προτάσεις σχετικά με τις μελλοντικέ εργασίες του φόρουμ. Ε, πρόκειται για προτάσεις που αφορούν ε, στη διαμόρφωση αυτής της ε, συνεργασίας. Η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει πολλά νέα στοιχεία. Αυτό που αναφέρεται κυρίως είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Τα περισσότερα προβλήματα αναφέρονται και στην ε, ανακοίνωση του 2006. Εδώ γίνεται λόγος για νέα προγράμματα σπουδών τα οποία θα πρέπει να προσανατολίζονται στο τι είναι χρήσιμο. Είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι γνώσεις ε, οι γνώσεις να μεταφερθούν στην πράξη. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, το προσωπικό των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων να μπορεί να μετακινηθεί με μεγαλύτερη ευκολία. Ε, σημασία έχει η περαιτέρω εκπαίδευση και η διακυβέρνηση για μια συνεργασία που είναι αποτελεσματικότερη. Όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι ήδη γνωστά και έχουν αναφερθεί σε παλαιότερα έγγραφα. Αυτό που είναι νέο και επίκαιρο τώρα πλέον είναι το τι πρόκειται να γίνει με μελλοντικές δράσεις. Και εδώ θεωρώ σημαντικό το εξής. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για νέες ε, μορφές ε, συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα αυτό ήταν επίμαχο. Τώρα, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί, αυτή η μορφή συνεργασίας βρίσκεται πάνω από προσωπικές ε, επαφές, πάνω από τη συμμετοχή σε σεμινάρια Αυτή οι μη δομημένες μορφές συνεργασίας ε, ίσως είναι αποτελεσματικότερες από τις ε, επίσημες δομές, οι οποίες επίσημες δομές ε, πολλές φορές είναι ιδιαίτερα περιοριστικές, άκαμπτες και τα πανεπιστήμια δεν έχουν μόνο την ε, αποστολή της ε, καινοτομίας αλλά ε, και καθήκοντα έρευνας και περαιτέρω κατάρτισης. Στην πρώτη πρόταση του εγγράφου που κατέθεσε η Κομισιόν αναφέρεται πολύ σωστά ότι οφείλουν τα πανεπιστήμια να προάγουν τις καινοτομίες, να βελτιώνουν τη γνώση γιατί είναι το κέντρο και η καρδιά του τριγώνου της γνώσης. Ενδέχεται λοιπόν αν ε, τελικά καταλήξουμε σε υπερβολικές ρυθμίσεις με αυτή, την, ε, τη μορφή να καταπνίξουμε την ευελιξία και να μην πετύχουμε το στόχο μας. Καλό είναι να υπάρχει διάλογος ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια και αυτό να επεκταθεί και στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια θαυμάσια πρόταση. Ε, βεβαίως, εφόσον ο διάλογος ε, γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ε, να επιβάλλει κανείς ε, στα πανεπιστήμια την επιχειρηματική σφραγίδα. Αντίθετα, το αντίθετο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή στις επιχειρήσεις να διεισδύσει η επιχειρηματική νοοτροπία. Να υπάρχει ένα είδος εταιρείας πανεπιστήμιο. Και εγώ συμφωνώ με την ε, Κομισιόν ότι στο πλαίσιο του διαλόγου ε, πρέπει και μπορούμε να εντοπίσουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις και να προσανατολιστούμε στο καλύτερο που μπορεί να υπάρξει τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο να ε, διευκολυνθεί μεταφορά γνώσης ανάμεσα στα ε, πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Τα πανεπιστήμια είναι ανοιχτά απέναντι σε κίνητρα που μπορούν να προκύψουν από ε, την περιφέρεια. Κύριε Πρόεδρε, Είπατε ότι πρέπει να είμαι σύντομη. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σταματήσω και βεβαίως είμαι ανοιχτή σε των συναδέλφων. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σύντομοι. όλα αυτά θα ακούσουμε δύο συναδέλφους. Να σας παρακαλέσω όμως να είστε πολύ σύντομοι. Μπάλσο και μετά η κυρία Ριέρα Μαδουρέλ. Ε, ευχαριστώ. πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι με αυτή την ανακοίνωση. Ε, υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και περί τίνος μιλάμε εδώ πέρα τώρα συγκεκριμένα είναι τα ενεργητικά, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, η ανταλλαγή ερευνητών μεταξύ των κρατών μελών, Μιλάμε για τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους εκπρόσωπους τους ε, βιομηχανίες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για έναν τομέα τον οποίο γνωρίζω εδώ και 34 χρόνια. Ήμουν 34 χρόνια ε, σε ένα πολυτεχνείο και η σχέση ε, μεταξύ των πανεπιστημίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ως εξή τουλάχιστον στο δικό μου πανεπιστήμιο. Όταν φτάσουν στο τελευταίο εξάμεινο οι φοιτητέ και γράφουν την πτυχιακή τους εργασία. Υπάρχει στενή συνεργασία με επιχειρήσεις μικρές και άλλες και είναι κάποιες μέρες σε μια επιχείρηση οι φοιτητέ και κάποιες μέρες στο πανεπιστήμιο και αυτό ωφελεί και την αγορά εργασίας και ε, το πανεπιστήμιο και οι εταιρείε ε, έχουν μετά άτομα τα οποία έχουν μια κάποια εμπειρία και βεβαίως ε, χρηματοδοτεί και η εταιρεία τις σπουδές και εξακολουθούν να παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι επαφές και μετά. Ε, μιλάμε λοιπόν για ποιοτική εκπαίδευση και σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, το, οι απόφοιτοι αυτοί κάνουν μετά και κάποιο διδακτορικό και εξακολουθούν να έχουν επαφές νομίζω τα ίδια ισχύουν και στην Δυτική ε, Ευρώπη ε, εγώ θεωρώ λοιπόν πως ε, μπορούμε να αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα αν είχαμε αυτές τις, τις περιόδους να επεκταθούν σε μια περίοδο δύο ετών. Παρακαλώ και εσείς σύντομοι Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η εκπροσώπηση των πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Θα έχουμε μία, ένα σημείο επαφή ή πολλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο εδώ πέρα. Υπάρχει ένα συμβούλιο πανεπιστημίων ε, και εγώ όταν έκανα μια έκθεση του 2000 ήταν η εκπρόσωπη των Πριτάνεων και όχι των πανεπιστημίων. Οπότε είναι οι Πριτάνης, οι κοσμήτορες που προσπαθούν ε, να περάσουν τα δικά τους. Εάν δείτε δε το τι γίνεται σε σχέση με την ε, αγορά εργασίας ε, δεν υπάρχει εκεί κάποια εκπροσώπηση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν νομίζω κάποια κριτήρια ε, ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων και την σύνδεση με τις επιχειρήσεις και μετά δείτε εδώ πέρα τι αναφέρεται στο, στο κείμενο. Ε, κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, οι επιχειρήσεις ε, χάνουν ε, από τις επενδύσεις τους στην έρευνα Οπότε γιατί να μην υπάρχει μια έκπτωση του ΦΠΑ για δύο-τρία χρόνια για να βοηθηθούν οι καινούριες ε, επιχειρήσεις. Για αλλιώς δεν θα βρούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειαζόμαστε για να καταβάλουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έρευνας ε, και ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία θα είναι και γενικότερη όσον αφορά την χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ και Καρβάλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Να σας πω πως ε, το έγγραφο αυτό εδώ πέρα της Κομισιόν δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Εγώ νόμιζα πως θα μπορούσαμε να βασιστούμε στην εμπειρία πολλών κρατών μελών ε, στον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων τους ε, δηλαδή πρέπει να συνδεθούν καλύτερα με τις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται και στη Γερμανία με τη σχετική πρωτοβουλία αριστείας και στη Γαλλία και δεν ξέρω, στην Κομισιόν θα μπορούσαν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας του EIT. Νομίζω πως η επόμενη γενιά προγραμμάτων θα πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να εξυγχρονιστεί το σύστημα όχι μόνο των πανεπιστημίων, πρέπει να εξυγχρονιστεί σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολο για τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και την, τις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή και πρέπει να αποτελέσει αν θέλετε έμβριο νέων κατευθυντήριων γραμμών για να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα στο Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συνοδελέφους ε, που είχαν 11 Ιανουαρίου υποβολή της έκθεσης, 27 Ιανουαρίου τροπολογίες, 22-23 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, 23 Μαρτίου στην Επιτροπή Πολιτισμού και τον Απρίλιο, αν όλα πάνε καλά, στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης και θα ήθελα να χαιρετήσω τον Γενικό ε, Διευθυντή τον εργαστά του Γενικού Διευθυντή κ. Δελμπέκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Κύριε Δελμπέκε, παρακαλώ. Σα καλωσορίζω, Σα ευχαριστώ που δείξατε κάποια υπομονή. Έχουμε καθυστέρηση χρονική, αλλά θέλουμε και αυτό το θέμα να το εξετάσουμε. Πρόκειται για την προπαρασκευαστική εργασία για την εφαρμογή του Σύμβουλου Εμπορίου Εκπομπών του ETS που μα απασχόλησε πέρσι πάρα πολύ. Η Αρμόδια Επιτροπή η Περιβάλλοντος ασχολείται ήδη έντονα με το θέμα και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την δυνατότητα να συζητήσουμε. Κύριε Τελμπέκη, έχετε το λόγο. Για πέστε μας πού βρίσκονται οι προκατορικές εργασίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση να είμαι εδώ και να σας παρουσιάσω κάποια πρόοδο που πετύχαμε στην εφαρμογή της οδηγίας για το σύστημα εμπορίου εκπομπών που υιοθετήθηκε πέρσι το Δεκέμβριο. Η αναθερωμένη οδηγία συμπεριλαμβάνει ε, μεγάλο ρυθμό μέτρων εφαρμοστικών. Το καθένα υπάρχει στην διαδικασία ε, εφαρμογής με εποπτεία. Έχει προωθήσει τις εργασίες οικομισιών και βρίσκεται ευθυγραμμασμένη με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στην οδηγία. Θα μου επιτρέψετε να τονίσω πέντε σημεία, πέντε μέτρα εφαρμοστικά. Το πρώτο είναι η διαρροή του, του άνθρακα. Το πρώτο μέτρο που περνάει είναι η έγκριση του καταλόγου των τομέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο για την διαρροή αυτή και επιτεύχθη τη 18 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλλαγή Κλίματο και το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή εξετάζει το λόγο κείμενο. Ο κατάλογος που προτάθη από την Επιτροπή για τις Κλιματολογικές Αλλαγές θα πρέπει να υιοθετηθεί σε περίπτωση κατά την οποία η δέσμη που έχει καθοριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2009 σε φασμού και αν όλα προχωρήσουν καλά και συμφωνήσει το Κοινοβούλιο, η έγκριση στην Κομισιόν προβλέπεται 22-23 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο κατάλογος ισχύει μέχρι 5 χρόνια και ενδεχομένω να πρέπει να προσθεθούν κάποια άλλοι εάν πληρούν ε, κάποια ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Θέλουμε να τονίσουμε επίσης ότι η απόφαση Ε, προβλέπει 20% ε, μείωση μονομερή και στην περίπτωση που άλλα κράτη δεν συμφωνήσουν για τη μείωση των δικών του εκπομπών. Είναι λοιπόν οπωσδήποτε αντικείμενο αναθεωρήσεις πριν από το 2014 υπό το φως του αποτελεσμάτων της συμφωνίας της ε, Κοπενχάγης. Δύο αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν. Το πρώτο είναι ότι ανάλογα από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν κάποια κράτη μπορεί να αλλάξουν τα στοιχεία εμπορίας. Και μέσα στα πλαίσια της συζήτησής μας για το benchmarking θα ξέρουμε καλύτερα πόσο ακριβώς δίδεται ανατομέα. Θα μου επιτρέψετε όμως να επαναλάβω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από 8-9 μέρες επιβεβαιώσε ότι ο κατάλογος που υπάρχει τώρα επιτάπτως ενώπιον ημών θα αναθεωρηθεί υπό το φως του αποτελέσματο των διαπραγματεύσεων διεθνώ για τι κλιματολογικέ αλλαγέ. Αν υπάρχουν αλλαγέ στον κατάλογο αυτό βασιζόμενε στη συμφωνία τη ε, Κοπενχάγη, οι αλλαγέ αυτέ θα αποφασιστούν από αυτό το Κοινοβούλιο μαζί και με το Συμβούλιο κατόπιν τη Κοπενχάγη. Αυτό είναι για το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι για το benchmarking έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια καθορισμού ε, φιλοδόξων και εναρμοσμένων κοινοτικών benchmark. Πολλοί από εσά είναι ισοδυνήμοροι ότι η προπαρασκευαστική εργασία προχωράει σωστά και ότι οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους λαμβάνουν χώρα. Το τρίτο τμήμα που θα ήθελα να τονίσω είναι η ε, δημοπράτηση. Η δημοπράτηση θα είναι η κύρια μέθοδος εμπορίας των εκπομπών αυτών. Και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του επόμενου έτους θα πρέπει να εορτηθεί ο σχετικός κανονισμός για τη δημοπράτηση. Και εκεί δηλαδή πραγματοποιούμε προπαρασκευαστικές εργασίες η γραπτή διαβούλευση των ενδιαφερομένων ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Τα αποτελέσματα της γραπτής αυτής διαβούλευσης έτυχαν επεξεργασία και συμπεριλαμβάνονται σε ένα σκιαγράφημα του κανονισμού που συζητιέται και πάλι με τους ενδιαφερόμενους. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή διατυπώνει τον κανονισμό της υπό το φως της υποβολής στην Επιτροπή για τι Κλιματολογικές Αλλαγές Γενάρη με Φλεβάρι του 2010 και μετά την υιοθέτησή του στην Επιτροπή αυτή θα υπάρχουν τρεις μήνες για εξέταση του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αυτό θα μας επιτρέψει να υιοθετηθεί ο κανονισμός από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2010 όπως προβλέπεται στην οδηγία. Το τέταρτο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η εργασία της Κομισιόν στην προστασία της αγοράς του άνθρακα κατά ε, παρατυπιών και καταχρήσεων της αγοράς. Η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσον η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ETS ε προστατεύεται επαρκώς από καταχρήσεις στην αγορά. Η Γενική Διεύθυνση Τρέν Περιβάλλοντος και Μάρκτ συνεργάζονται στενά για να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και εμείς μελετάμε και παρακολουθούμε στενά σχετικές συζητήσεις και στο Αμερικανικό Κογκρέσο για το θέμα αυτό. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την επιτήρηση της αγοράς και θα είναι κατά πάσα φαινότητα τμήμα μελλοντικής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Η εκτελεστική περιοχή θα πρέπει να σας κάνει μια έκθεση για το θέμα αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους και όποια νομοθετική πρόταση θεωρεί η Κομισιόν χρήσιμη θα πρέπει να περάσει από την πλήρη διαδικασία στην Το πέμπτο και τελευταίο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η εργασία που ολοκληρώνει η Κομισιόν όσον αφορά την συλλογή και αποθήκευση του άνθρακα. Γιατί θα θυμόσαστε ότι υπάρχουν 350 εκατομμύρια άδειε που έχουν τεθεί κατά μέλλον. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα 450 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά η ανάπτυξη του CCS θεωρούμε ότι είναι μια καλή δυνατότητα που μπορεί να αναπτυχθεί στο, για το μέλλον. Και η Κομισιόν προτίθεται τις επόμενες εβδομάδες να τελειοποιήσει το σχέδιο και να υποβάλει στην Επιτροπή Κραματολογικών Αναγών την πρόταση αυτή, ίσω όχι πριν από τα τέλη του έτου, αλλά οπωσδήποτε αμέσω μετά την αρχή του καινούργιου έτου. Θέλουμε να προτείνουμε μια κοινή κοινοτική προσέγγιση που θα εξισορροπεί γεωγραφικές και τεχνολογικές εξελίξεις και επίσης με έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να τονίσω. Υπάρχουν και άλλα πολλά διαφορετικά θέματα που θα μπορούσα να σας παρουσιάσω. Αυτά όμως είναι τα πέντε πιο σημαντικά θέματα που έχουμε ενώπιον ημών μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας και εν το χρόνο θα σας υποβάλλουμε και άλλες προτάσεις. Αλλά τα πέντε σημεία που τόνισα είναι εκείνα που οδηγούν σε περισσότερο ενδιαφέρον και του σώματός σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κλιματολογικά θέματα και ήθελα να τονίσω τα πέντε αυτά θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να ε, ακολουθήσει το πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που μας επιβλήθη. Αλλά πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι ε, συμμετέχει αυτή η Επιτροπή. Πάντως, ε, η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος νομίζω ότι είναι η μόνη αρμόδια επί του θέματος. Όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε και εμείς. Το είχαμε συμφωνήσει ευθύς εξ αρχής. Και όταν μιλάτε για ε, κλιματική αλλαγή, ε, φαντάζομαι η Επιτροπή για το Κλίμα, φαντάζομαι εννοούστε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όχι μια νέα Επιτροπή, υποσύσταση. Η συνάδελφος κυρία Νίπλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, καλωσορίζουμε στην Επιτροπή ε, και για ε, το ότι θελήσατε να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς ισχύει στην οδηγία περί ανταλλαγής ποσοστώσεων για τις εκπομπές. Όσον αφορά το τελευταίο θέμα που είπατε, θέλω να τοποθετηθώ επ' αυτού για τα 300 εκατομμύρια για, το, για την δέσμευση ε, και την αποθήκευση του άνθρακα και για νέα προγράμματα ενέργειας. Αυτά θα αφαιρεθούν από το απόθεμα. Έτσι το είχαμε συμφωνήσει. Εγώ όμως ρωτώ συγκεκριμένα, ποιος θα αποφασίσει για αυτά τα προγράμματα τα οποία υποτίθεται θα χρησιμοποιηθούν από το απόθεμα των 300 εκατομμυρίων. Και ποιο ορίζει ποια προγράμματα είναι καινοτόμα, ποια όχι. Και πώς γίνεται η κατανομή ανάμεσα στα προγράμματα CCS και αυτά για, την, ε, για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Εμένα με ενδιαφέρει να γνωρίζω πώς λαμβάνονται οι αποφάσει ε, και στη τελική ανάλυση ε, ποιο τι παίρνει τις αποφάσεις. Δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξή. Exposed Carbon Leakage List. Και το είπατε κι εσείς, ε, αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο γίνονται οι σχετικές έρευνες και Υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση στα πολωνικά. Εντάξει. Λοιπόν, Τώρα, όσον αφορά αυτό τον κατάλογο, είπατε ότι το 2014 θα έχουμε αναθεώρηση έχοντας κατά νου και το τι ακριβώς ε, προσδοκούμε από την Κοπεχάγη στο τέλος του έτους. Ερωτώ λοιπόν, εσείς στις προετοιμασίες για την Κοπεχάγη συμμετέχετε ή όχι. Και με ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη, δηλαδή τελικά τι πιστεύετε εσείς ότι θα προκύψει από την Κοπενχάγη. Εντάξει, ξέρω ότι δεν μπορείτε να λάβετε επίσημη θέση, όμως με ενδιαφέρει η προσωπική σας. Φαντάζομαι θα συμμετέχετε στις διαδικασίες, φαντάζομαι έχετε επαφές και με τους Αμερικανούς. Θα ήθελα να γνωρίζω εσείς κατά τη γνώμη σας το τέλος του έτους τι θα προκύψει από την Κοπεχάγη. Και έχω και μία ερώτηση. Δηλαδή, την τελευταία φορά στην Ολομέλεια ε, ακούσαμε τον Επίτροπο για ε, την Ενέργεια, αρμόδιο και για το πρόγραμμα Desertic, ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την Ευρώπη. Και το ερώτημά μου κατά πόσον ε, το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δηλαδή, ε, μήπως υπάρχουν σκέψεις στα πιστοποιητικά εκπομπών ότι υπολογιστεί στο πρόγραμμα της να προσμετράτε και στο πρόγραμμα της Κομισιόν. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια καλή σκέψη για να δοθούν κίνητρα και ερωτώ. Έχετε σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο ε, πρόγραμμα των πιστοποιητικών εκπομπών, επειδή αναφέρεται ε, στο πρόγραμμά μας, αλλά ίσως υπάρχουν και άλλες σκέψεις να δοθούν κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία να συμμετάσχει και αυτή σε αυτά τα προγράμματα. Και τελευταία παρατήρηση προς τον πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είπατε ότι η Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, που το επισημάνατε. Παρακαλώ να διευκρινίσετε για άλλη μια φορά ότι η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Ενέργειας, που συμμετείχε παλαιότερα σε θέματα κλιματικών αλλαγών, να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά με τη συνεργασία ή με άλλα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως Επιτροπή Βιομηχανίας να συνεχίσουμε να αφήνουμε τη σφραγίδα μας. Και Εγώ σας ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες. Μια παρατήρηση πρώτα, εάν μου επιτρέπετε, που αφορά την επιστήμη. Πολλοί ερευνητές, ε, όλο και περισσότεροι στη Γερμανία, ερευνητές έχουν κάποιες αμφιβολίες, γιατί εδώ και δέκα χρόνια παραμένει σταθερή και μειώνεται η θερμοκρασία της γης. Και αυτό είναι η προβλέψη για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, ότι θα μειώνει θερμοκρασία παρά τις αυξημένες εκπομπές. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν ε, αυτά τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν φτάσει στην Κομισιόν και ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε. Πρώτο ερώτημα. Κατόπιν εκπλήσωμε κάπως για το δεσμευτικό πρόγραμμα που έχετε εδώ πέρα υποβάλει μέχρι τον Ιανουάριο Φεβρουάριο του 2010 και πρέπει να παρουσιαστούν ε, όλα αυτά στην Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής που ευτυχώς βεβαίως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν θυμάμαι καλά, ολόκληρο το πακέτο ETS ε, ήταν υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας στην Κοπενχάγη και ήταν νομίζω και ζήτημα το να συμφωνήσουμε στα βασικά στην Κοπενχάγη και δεν είναι καθόλου αυτονόητο η δε Γερμανίδα Καγκελάριος που συγκινείται πάρα πολύ ε, με την κλιματική αλλαγή μιλάει πλέον μόνο για μία συμφωνία πλαίσιο και όχι για δεσμευτικούς στόχους πλέον στην ε, ε, Κοπενχάγη. Σας αρκεί εσάς μια συμφωνία πλαίσιο για να οδηγηθείτε σε υποχρεωτικό σύστημα πληστηριασμού εάν δεν συμφωνήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα ήθελα λοιπόν να έχω σαφείς πληροφορίες, μήπως έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση στην οποία πραγματικά καταλήξουμε μόνο σε μια συμφωνία πλαίσιο. Τελευταία ερώτηση, Τίκαου και μετά θα ακούσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ομιλητή μας για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Το δε πακέτο ενέργειας κλίματος ε, δεν αφορά μόνο το ETS, αφορά και την δέσμευση των κρατών μελών να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Στο δε πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την χρηματοδότηση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, γιατί ε, οι σχετικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν δυσκολία σήμερα να βρουν την χρηματοδότηση τους πόρους για να εξυγχρονιστούν για να μπορέσουν με τη σειρά τους ε, να συνεχίσουν να παράγουν αλλά με χαμηλότερες εκπομπές. Και επίσης με τον τομέα που θα μείνει εκτός της εμπορίας, δηλαδή τομέας ε, μεταφορών και κτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων ζήτησε να έχουμε περισσότερους πόρους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Και Ελπίζω για την επόμενη προγραμματική περίοδο να μας βοηθήσετε να αυξήσουμε την ποσόστοση από το Ταμείο ΦΕΝΤΕΡ για να ξοδέψουμε περισσότερα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντελμπέκε τώρα έχει να απαντήσει σε ένα ολόκληρο πακέτο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Είναι ένα γενικό ερώτημα ε, στο οποίο θα ήθελα να αφιερώσω λίγες στιγμές για το πιθανό αποτέλεσμα της Κοπενχάγης και το ρώτησαν αρκετοί. Πράγματι η Κοπενχάγη μάλλον δεν θα καταλήξει σε μια συνθήκη διάδοχο του πρωτοκόλλου του Κιώτο που θα έχει δεσμευτικούς στόχους. Θα έχουμε πολιτική συμφωνία γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει πως οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία πρέπει να είναι δεσμευτική στην Κοπενχάγη και αμέσως μετά πρέπει να εξειδικευτεί σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο. Οπότε θα συνεχιστεί η δουλειά και μετά την Κοπενχάγη και δεν έχει κρυθεί ακόμα το εάν θα έχουμε ε, μία σύνοδο τρει ή έξι μήνες μετά την Κομπεχάγη. Αυτό θα γίνει πριν από την πρώτη κοπ του χρόνου το Δεκέμβριο στο Μεξικό. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε εγκαταλείψει την ιδέα μιας δεσμευτικής συνθήκης γιατί η συνθήκη της Κομεχάγης πρέπει να αποτελέσει διαδοχό του Κιώτο. Ποια στοιχεία τώρα αναμένουμε στη συμφωνία της ε, Κοπενχάγης. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε σημαντικά στοιχεία θα πρέπει να εμφανιστούν. Το πρώτο είναι η μείωση των εκπομπών. Δεν βλέπω πως δεν θα συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο στην Κοπενχάγη και εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσουμε επιτυχία. Γιατί θέλουμε μείωση από τις ανεπτυγμένες χώρες από 25 έως 40% αλλά θέλουμε και απτές μειώσεις οι δράσεις τέτοιες από τις ανερχόμενες οικονομίες. 15-30% από τα συνήθεια έχουμε πει. Νομίζω το μήνυμα αυτό έχει ληφθεί. Η Κίνα και η Ινδία μάλλον προς τα εκεί πηγαίνουν. Οπότε μείωση των εκπομπών θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο και Αναμένουμε βεβαίως ε, μειώσεις και από τις ε, ανεπτυγμένες χώρες, ήπα ε, και από τις αναπτυσσόμενες Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική κλπ. Τα άλλα στοιχεία αφορούν τεχνολογία, με τη δέσμευση κτλ, προσαρμογή, αποδάσωση και θα είναι ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας. κατόπιν το ερώτημα του κυρίου Πίπερ. Ε, αλλάζουμε τώρα οτιδήποτε ευθύθηκε πέρσι στο πακέτο ενέργειας και κλίματος. Το ETS, η οδηγία CCS, όλα αυτά αποτελούν μία μονομερή ε, δέσμευση για μείωση μέχρι 20% μέχρι το 2020 ε, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Πρόκειται για μονομερή δέσμευση. Είπε η Ευρώπη ότι θα μπορούμε το 20% να το κάνουμε και 30% εάν ε, στην Κοπενχάγη οι λοιπές χώρες ε, επίσης αναλάβουν να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες. Οπότε το 20% είναι ήδη νομοθεσία και το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής ε, έχει οριστεί από τον νομοθέτη οριστεί μεγάλη λεπτομέρεια. Όλοι δυσκολευόμαστε και το ETS ε, καθώς έχει σχεδιαστεί για την περίοδο 2013-2020 εξακολουθεί να ισχύει όπως συμφωνήθηκε πέρσι τον Νοέμβρη. Τώρα με ρωτήσετε αν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο. Ε, το εναλλακτικό σχέδιο θα τεθεί στην Κοπεχάγη και αμέσως μετά, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν και οι άλλοι. Η Ευρώπη θα αναθεωρήσει το στόχο της 30% και πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει με το... με το να μοιράσουμε την προσπάθεια, με τις προσπάθειες δασοκομείας κτλ. Και τα τρία τελευταία αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή το RED, ε, ζητήματα αποδάσωσης, ε, αλλαγή χρήσης γης ε, και δασοκομεία στην Ευρώπη δεν αποτελούν μέρος της μονομερούς δέσμευσης 20% και μπορούν να αποτελέσουν μια συνέχεια της, συμφωνία της συμφωνίας στην Κοπενχάγη. Κατόπιν ένα συγκεκριμένο ερώτημα της κυρίας Νίμπλερ για το πώς θα οριστούν τα 300 εκατομμύρια που θα μπουν σε ένα απόθεμα, Ποιο αποφασίζει το τέλος. Θεωρούμε ότι θα γίνει σε δύο τμήματα η απόφαση. Έχουμε ένα σχέδιο απόφασης που θα πρέπει να ενσωματώνει όλα τα βασικά στοιχεία του πώ θα διατεθούν τα 400 εκατομμύρια. Μιλάμε για το ότι θα μοιραστούν την κατανομή στο χαρτοφυλάκιο το τεχνολογικό, την κατανομή στα κράτη-μέλη, ποιος θα κάνει την ανάλυση, Όλα αυτά πρέπει να περιγραφούν σε αυτή την απόφαση. Και πρέπει να κάνουν εδώ πέρα σοβαρή δουλειά και τα κρατημέλη, γιατί πρέπει να κάνουν την προεπιλογή των έργων που θα φέρουν για την εκταμίευση των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση, είναι διαδικασία επιτροπολογίας αλλά θεωρώ πως υπάρχει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ πέρα να παίξουν τα κρατημέλη και εμεί θέλουμε πλήρη δέσμευση των κρατών μελών και εμπλοκή. Κατόπιν το Desert Tech για το εάν θα μπορεί να επιλεγεί. Μπορεί να είναι επιλέξιμο για πιστώσεις εμπορίας, αλλά όχι για το αποθεματικό, γιατί αυτό πάει μόνο για έργα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το Desert Tech φαντάζομαι θα είναι στην έρημο, οπότε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσο έχουμε ε, δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό για τις, ε, τους νέους ερχόμενους, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, κονδύλια RTD, CTM, ακόμα και διαρθρωτικών ταμείων ε, ή ταμείου συνοχής, ε, τα κονδύλια στο μέτρο που είναι διαθέσιμα για τρίτες χώρες. Μετά υπήρχε ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τις τελευταίες εξελίξεις στα επιστημονικά δεδομένα. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε. Βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ σε αυτά τα οποία λέει το IPPC, το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή και καθώς το IPPC ε, μας δίνει τις κατευθύνσεις, το IPPC πρέπει πρώτα να εξετάσει το πάνελ αυτό, ε, τα στοιχεία αυτά. Ακούω πως υπάρχουν νέα στοιχεία, πως η θερμοκρασία σταθεροποιείται. Άλλοι λένε πως τα 450 μέρη στο εκατομμύριο το βασικό σενάριο είναι πολύ χαλαρό, πως πρέπει να το κάνουμε ακόμη πιο αυστηρό. Αντιστεκόμαστε και σε αυτές τις ε, απόπειρες, γιατί θέλουμε να βασιστούμε στην συνένεση, ας πούμε, της ε, κοινότητας ε, της επιστημονικής και είμαστε καταδικασμένοι νομίζω να αναμένουμε να περάσει αυτή η πιθανή αλλαγή των κλιματικών δομένων από το IPPC. Υπάρχει σχέδιο για το 2014 νομίζω προβλέπεται μια επανεξέταση, αλλά πάντα προβλέπονται πιθανές αναθεωρήσεις. Μετά είχαμε το ερώτημα της κυρίας Τικάου για την χρήση χρηματοδότησης για την εσωτερική προσαρμογή και μείωση των επιπτώσεων εντός της Ευρώπης ελπίζω στο τελευταίο έγγραφο, στην τελευταία ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του κλίματος, η Κομισιόν προτείνει σαφώς να αναλυφθούν περισσότερες δράσεις και να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και ελπίζω στην συζήτηση των δημοσιονομικών προοπτικών ε, που θα ακολουθεί στα επόμενα χρόνια να είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Πώς δηλαδή τα χρήματα αυτά θα έρθουν πιο κοντά στους στόχους πολιτικής της Ένωσης. Οπότε αυτό οπωσδήποτε ισχύει για τα κτίρια, για τις μεταφορές. Να υποστηρίξουμε αυτές τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της οδηγίας του να μοιραστεί ο φόρτος. Τώρα όσον αφορά τις εταιρείες, οι εταιρείες καλύπτονται από το ETS. Το πρόγραμμα νομίζω είναι αρκετά αυστηρό μέχρι το 2012. Από το 2013 έχουμε το νέο καθεστώς εμπορίας και οποιαδήποτε δημόσια στήριξη προς τις εταιρείες του ETS πρέπει να περάσει α, βεβαίως και την βάσανο των διατάξεων κρατικών ενισχύσεων. Εάν λοιπόν αυτές οι διατάξεις γίνουν σεβαστές δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι η βασική χρηματοδότηση των εταιρεών και ελπίζουμε πως η αγορά διοξιδίου του άνθρακα θα ανταμείψει τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών. Και αυτό το οποίο παρατήρησα ειδικά και στα νέα κράτη-μέλη που χτίζουν καινούριο τομέα ενέργειας ε, είναι ήδη ενσωματωμένη η τεχνολογία χαμηλών εκπομπών στον τομέα της ενέργειας. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ε, να δεχτώ και άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέντε έχουν σβήσει ακόμα το λόγο. Πέντε λεπτά έχουμε στη διάθεσή μα. Ο καθένα, παρακαλώ ένα λεπτό για να προφτάσει και η Κομισιόν να απαντήσει. Ο κ. Ζαλό. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα το ότι ελέγχθη ότι μετά την Κοπεχάγη ενδεχομένω θα αναθεωρηθεί ο κατάλογος. Έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν για το θέμα του benchmarking. Η Κομισιόν θα διατηρήσει τον κανόνα που αναφέρεται στην οδηγία για το ΙΤΕΣ, δηλαδή το benchmark στο 10% των πιο αποτελεσματικών εγκαταστάσεων. Αυτό δεν το αναφέρατε καθόλου υπάρχει έντονη πίεση να πολυπλασιαστούν οι ορισμοί για το benchmarking και ίσως τελικά αυτό που δυναμώσει την οδηγία. Δεύτερον, συσχετίσατε τις ε, διαρροές ε, άνθρακα και το θέμα των δωρεάν ε, χορηγήσεων. Κάνει κάτι σχετικά η Κομισιόν. Γιατί σήμερα μπορεί μια εταιρεία να ε, μετατοπίσει την παραγωγή της και παρόλα αυτά να έχει δικαίωμα σε δωρεάν ποσοστώσεις. Μετά είπατε δεν υπάρχει καμία δέσμευση για άλλε χώρε εκτό από τις χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί όμω είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Ντεμπόρ και μα είπε ότι και άλλε χώρε αυτή τη στιγμή αναλαμβάνουν σημαντικέ δεσμεύσει. Και στον ορισμό του καταλόγου του τομέα που θα ωφεληθούν από παρεκκλήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη οι δεσμεύσει άλλων κρατών. Και δεν μπορούμε να εξακολουθούμε να προσποιούμεθα ότι η Ευρώπη είναι η μόνη στον κόσμο που καταβάλει προσπάθειες. Τέλος, βλέπουμε ότι με την οικονομική κρίση υπάρχει πτώση των εκπομπών. Και αυτό που λένε οι οικονομολόγοι είναι ότι σήμερα η προσπάθεια για να πετευχθεί το 30% της μείωσης ε, των εκπομπών παρά τις προσπάθειες που προβλέπονται πριν από ένα χρόνια για να επιτευχθεί μια μείωση των εκπομπών του 20%. Από την άλλη μεριά ακούμε στην Ελληνική Διεύθυνση Περιβάλλον, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεται αυτό, ότι τέλος ένας περιοριστικός στόχος του μείωσης του 20% για την κατανάλωση της ενέργειας, όπως είπε και η κυρία Τικάου, θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο για την αγορά άνθρακα, γιατί αυτό θα μείωνε συνεχώς την τιμή ανατών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες ασυνέπειες που υπάρχουν σε αυτό που μας λέει η Κομισιόν και θα θέλαμε να υπάρχει περισσότερη συνοχή και περισσότερη φιλοδοξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος και ο Σβόγγεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στην Ουαλία έχουμε πολλά αποθέματα άνθρακα, γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, ε, το μέλλον ε, των ανθρακοριχείων στην Ουαλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την εξέλιξη του CCS. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε τέσσερα πιλωτικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχα κάποιες ε, ερωτήσεις σχετικά με τα χρήματα που θα ε, διατεθούν. Είπατε ότι θα υπάρξει κριτήριο γεωγραφικό αλλά και κριτήριο τεχνολογίας. Τώρα, όσον αφορά τη τεχνολογία, σε αυτή τη φάση η Κομισιόν προτιμάει κάποια ε, τεχνολογία προ ε, καύση, κατά διάρκεια της καύσης και μετά την καύση. Έχει κάποια προτίμηση. Κυρία. Κυρία Σκουρτίνες, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η έρευνα των τελευταίων ετών απέδειξε ότι το θέμα της, ε, του κλίματος είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εξελίσσεται τελείως διαφορετικά το κλίμα στο βορρά και αλλιώς στο νότο. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλοί δεν ε, λαμβάνουν υπόψη τους αυτή τη ε, διαφορά, τη διαφοροποίηση μεταξύ βορρά και νότου. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να μην σε αφήνεις. Το 20% των εκπομπών προέρχεται από τη βιομηχανία. Αυτό θα τεθεί υπόψη στην Κοπενχάγη. Η ε, γεωργία που παράγει όμως και αυτή η του άνθρακα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την επιδείνωση του κλίματος. Ε, δεν ε, έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικά θέμα. Βεβαίως, όταν μιλάει κανείς για τη γεωργία είναι σαν να πατάει πάνω σε αναμένα κάρβουνα η αλήθεια είναι η έρευνα δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ έτσι ώστε να μας δώσει κάποιες λύσεις για τα προβλήματα που προκαλούνται από τη Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Ε, συνεργαστήκαμε για πάρα πολλά χρόνια, ε, πρώτα στο Συμβούλιο και μετά στην Επιτροπή. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ε, κάτι που το υπογράμμισαν ήδη οι συνάδελφοί μου. Η Επιτροπή Βιομηχανίας είναι και Επιτροπή Αρμόδια για το Κλίμα και είχαμε μεγάλη επιτυχία στα θέματα της κλιματικής αλλαγής γιατί η Ευρώπη ε, διαπίστωσε ότι η στρατηγική είναι ένα ε, καθοριστικό χαρακτηριστικό του κλίματος και αυτό το χαρακτηριστικό μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνία και σήμερα να έχουμε μια θέση για την Κοπεχάγη. Έχω ένα ερώτημα σχετικά με τον άνθρακα, δέσμευση και αποθήκευση. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν περίπου 11 τέτοια προγράμματα, άνθρακα CCS και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Όμως το πρόγραμμα αποκατάστασης, εξ όσων γνωρίζω, στηρίζει μόνο την πρώτη φάση του κόστους για αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά πρόκειται να ε, χρηματοδοτηθούν ε, από τα 300 εκατομμύρια και αν ναι, πώς θα γίνει η ένταξη αυτών των προγραμμάτων σε 300 εκατομμύρια, τη στιγμή που υπάρχουν ήδη άλλες προτεραιότητες. Ο κύριος Πίμπα. Πολύ σύντομα, θα ήθελα να προ... Θέσω μία ερώτηση στις πολλές που σας υπευλήθησαν. Αναφέρεται στην πραγματική στην πραγματική πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος για Ανταλλαγή Ποσοστώσεων υπάρχει ένα πρόβλημα ορισμένε χώρες που παρεμποδίζουν ε, την απόφαση στο Συμβούλιο ε, προβλέπουν ε, να υπάρχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή. Κατά περίπτωση, η Κομισιόν δικαίως θεωρώ Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα, γιατί αυτό είναι πιο συνεπές, ορθολογιστικό και πιο οικονομικό. Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το σύστημα οργάνωσης στο οποίο θα καταλήξουμε. Μια που κάπως ε, αισιόδοξα θεωρούμε ότι η Κοπενχάγη θα είναι επιτυχία, ίσως όχι άμεσα, αλλά μακροπρόθεσμα. Και τι θα γίνει με αυτό το σύστημα περιορισμού και ποσοστώσεων. Ευχαριστώ κύριε Βίμπερ. Ο κ. Δεντέκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα του benchmarking, το σε ποιο βαθμό ε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη της οικομισιόν, το 10%. Το λαμβάνουμε σοβαρά, αλλά υπάρχει και δουλειά που έκανε ο νομοθέτης που είπε ότι το 10% θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως το σημείο αναφοράς για τη σύγκριση, για το benchmarking. Είναι λοιπόν ένα ε, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό η συζήτηση για το benchmarking αλλά ως ε, σημείο ε, κίνησης υπάρχει το 10% και όπως σας είπα αυτό συζητάμε με τη βιομηχανία. Στη τελική ανάλυση στο 10% ο σημείο κίνησης, εκεί υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή το σύνολο των ε, επιδοτήσεων ποσοτικά είναι περιορισμένο. Όσο πιο πολύ δίνει κανείς τον ένα, τόσο λιγότερα απομένουν για τον άλλο. Αυτό δεν έχει γίνει απόλυτα συνειδητό από όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τώρα, όσον αφορά το κόστος 20%, 30% ο στόχος πράγματι έχει ε, κατέβει προς τα κάτω με την ε, ύφεση μειώνονται οι εκπομπές καθότι υπάρχει λιγότερη οικονομική δραστηριότητα και ίσως αυτό να απαιτεί από εμά να, ε, να λαμβάνουμε λιγότερες ενέργειες. Και ναι και όχι. Η γραμμή της Κομισιόν είναι ότι έχει συμφωνηθεί η νομοθεσία για το 20% και οτιδήποτε πάνω από το 20% αυτό ε, θα είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί μετά την Κοπεχάγη. Η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει μελέτη αξιολόγησης, να κοινοποιήσει τα στοιχεία είμαι σίγουρος ότι αν τελικά η οικονομική δραστηριότητα δεν αναπτυχθεί όπως κατά το παρελθόν, τότε πράγματι θα μειωθεί το κόστος επίτευξης των στόχων που έχει θέσει ο νομοθέτης. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, ε, κατά πόσον η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει κάποια αίσθηση σχετικά με αυτό, θέλω να σας πω ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το τρίτο βασικότερο στοιχείο. Δηλαδή έχουμε στόχο για καινοτόμες ε, ενέργειες, ε, κατόπιν για τις εκπομπές και τέλος υπάρχει και το στοιχείο, το κριτήριο της απόδοσης, 20%, το οποίο ακόμα δεν έχει λάβει νομοθετική μορφή και αυτή είναι η διαφορά αφορά ε, της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο όμως οδηγούν το όλο σύστημα σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και ένα από τα βασικότερα στοιχεία του ETS ε, είναι ότι έχουμε σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα επενδυτικά μοντέλα των εταιριών. Ως εκ τούτου πρέπει λιγάκι να δούμε πώς όλα τα στοιχεία επιδρούν το ένα στο άλλο. Ε, έγινε μια ερώτηση σχετικά με την τεχνολογία CCT ε, αναφέρεται τρεις, αυτές όμως οι τρεις μπορούν να συνδυαστούν. Και είναι τη δέσμευση. Πρέπει να υπάρχει και αποθήκευση. Γι' αυτό εμείς αναμειγνύουμε τις ε, διάφορες ε, τεχνικές με τις διάφορες δυνατότητες αποθήκευσης. Έχουμε οκτώ κατηγορίες CCS και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια διεύρυνση. Πάντως η Κομισιόν, αν εσείς θέλετε να είναι 7-9, εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Τώρα, για την ερώτηση της κυρίας Κιουτέρες. Κοιτάξτε, η Γεωργία βεβαίως και είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και γίνονται πολλές ε, συζητήσεις ε, για την δασοπονία και για τη χρήση της γης. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη των στόχων, κυρίως αυτών που θα συμφωνηθούν στην Κοπεχάγη. Όσον αφορά τον έλεγχο, την αναφορά και την επαλήθευση, ακόμα δεν γνωρίζουμε με απόλυτη σαφήνεια τι θα συμβεί στην γεωργία σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε για τη βιομηχανία. Γι' αυτό και προς το παρόν διαφοροποιούμε την αγορά του άνθρακα από γεωργικές δραστηριότητες. Ερώτηση της κυρίας Καρβάλιο για τα προγράμματα CCS κατά πόσον ε, η υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Ανάκαμψης ε, μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα. Είναι δυνατόν γιατί τα προγράμματα CCS και η τεχνολογία είναι τόσο δαπανηρή που αν υπάρξει κάποιο συνδυασμός αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείε να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Ε, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κονδύλι για κάθε πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν οι ε, επικεφαλής, οι αρμόδιοι έχουν διαλέξει τουλάχιστον τρία ε, προγράμματα επίδειξης που επιτρέπουν το συνδυασμό. Και όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Βίμπα για να υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρατήσεων ή ε, το να πάνε προς τα εκεί τα αυτή είναι η άποψη της Κομισιόν, κατηγορηματικά, ότι χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα δημοπρατήσεων. Αυτό είναι το πιο λογικό που μπορεί να γίνει. Παρατήρησα βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εξηγήσει που πρέπει να δοθούν. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες ε, διοχετεύονται στα κράτη-μέλη και έτσι κάποια κράτη-μέλη ε, ξέρουν ότι αν δεν κάνουν τα ίδια τις δημοπρασίες θα έχουν ε, κάποια έσοδα. Εμείς λέμε στα κράτη-μέλη ότι στην περίπτωση που επιτρέψουμε διάφορες πλατφόρμες δημοπρασίες, αυτό θα είναι δαπανήρο και δεν θα αποτελεί καλή λύση για την Ευρώπη. Λέμε όμως επίσης ότι πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσει. Και υπάρχουν και ενδιάμεσες λύσεις ανάμεσα σε μια ε, ενιαία πλατφόρμα και διάφορες μπορούμε να έχουμε ένα υβριδικό σύστημα όπου η